συζητήσεις της συναδέλφου Τόια ακυρώνονται για σήμερα. Θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της 18 και 19 Ιουνίου. Τα σημεία λοιπόν 12, 13 και 14 δεν θα εξεταστούν σε αυτή τη συνεδρίαση. Το σημείο 20, τα σημεία 22 και 23 των συναδέλφων Μπάλτη και Γκίρκ θα αντιστραφούν το ένα στη θέση του άλλου και το σημείο 25 Καθώς ε, απουσιάζει ο συνάδελφος Μπόλτ, θα παρουσιαστεί από τον συνάδελφο Ποτόσνικ. Έχουμε διερμηνία. για όλες και προς όλες τις γλώσσες εκτός από ρουμανικά που θα έχουμε μόνο την για την που δεν θα έχουμε την πέμπτο πρωί και υπάρχουν αίθουσε ακροάσεων. Ξεκινάμε λοιπόν τις εργασίες της ε, συνάντησής μας. Ξεκινάμε με την ε, έκθεση του συναδέλφου Κορέη Αντεκάμπος για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, κύριε Κάμπος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα καλημέρα σε όλους. Ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους ε, συναδέλφους, τους κοιόδες συζητητές. Σας ευχαριστώ για τη σημαντική συμβολή που παρήχατε, για την ανταλλαγή απόψεων. Έγιναν πολλές ανταλλαγές απόψεων. Σας ευχαριστώ επίσης για το πνεύμα συνεργασίας ε, που επιδείξατε. Ήθελα να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες ε, και συνεισέφεραν με μεγάλο ενθουσιασμό, με πάρα πολλές ε, τροπολογίες, με στόχο τη βελτίωση, την τελειοποίηση αυτού του νομοθετικού σχεδίου. Ελπίζω ότι θα εξακολουθήσουν να δείχνουν ενδιαφέρον για το ζήτημα και στους μελλοντικού μας ε, διαλόγους είναι σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός, μιας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ακολουθήσει τα κράτη-μέλη αυτόνομα τις ενεργειακές πολιτικές χωρίς συντονισμένες επενδύσεις για την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών. Η καθαρή, φθηνή ενέργεια για τους πολίτες και τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι ακόμα μακριά εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγάλες προκλήσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως αυτό που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα με αυτή την ατομική προσέγγιση ήταν πολύ λίγο. Ό,τι έχει επιτευχθεί, έχει επιτευχθεί με ελλείψεις. Υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από τρίτες χώρες, υπήρξαν περιπτώσεις διακοπών των προμηθειών, ορισμένες γεωγραφικές περιοχές ε, δεν είναι καλά συνδεδεμένες. Υπάρχει ένας, ε, έχουμε μια αγορά όπου τα μέσα διασύνδεσης που υπάρχουν για το 2010 για το 10% ο στόχος του 10% δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ κρατών μελών έχει αυξηθεί κατά παραπάνω από το μισό την τελευταία δεκαετία σε σχέση με την προηγούμενη. Οι τιμές του φυσικού αερίου διαφέρουν ε, στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό γιατί σε ορισμένες χώρες υπάρχει υγροποιημένο αέριο σε χαμηλή τιμή που δεν φτάνει όμως σε όλα τις περιοχές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν μονοπωλιακές, ε, χαμηλής απόδοσης τοπικές αγορές, οι διασυνδέσεις δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν υπάρχει ελάχιστος ανταγωνισμός καθώς και ελάχιστα κίνητρα για να ε, πραγματοποιηθούν διασύνδεσεις. Το τίμημα που καταβάλει ο Ευρωπαίος καταναλωτής ε, για μια αποκλειστικά εθνική ενεργειακή υπηρεσία είναι πολύ υψηλό. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με τρόπο πιο ευρωπαϊκό για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά με ασφάλεια προμηθειών, ενεργειακή βιωσιμότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Για αυτό το σκοπό οι υποδομές ε, διασύνδεσης στην Ευρώπη είναι απαραίτητες και πρέπει να επιταχύνουμε την οικοδόμηση αυτών των υποδομών. Αυτός είναι ο ζωτικός στόχος του κανονισμού δεν πρόκειται λοιπόν για μια θεωρητική άσκηση για να εντοπίσουμε τα έργα προτεραιότητα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε παρουσιάσει τροπολογίες για την πρόταση της Κομισιόν με στόχο να δοθεί πιο ευρωπαϊκή χρειά στην όλη προσέγγιση, με, ε, μεγαλύτερο άνοιγμα και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων διαχειριστών. Το γεγονός ότι ε, εθνικά συμφέροντα μπορεί να μπλοκάρουν αυτές τις πρωτοβουλίες δεν είναι θετικό. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε αυτή τη στάση. Αντιθέτως θα πρέπει να επενδύσουμε σε έργα κοινού ενδιαφέροντος ή διαφορετικά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο, να αποφύγουμε τα κόστη κατασκευής να διωγγώνονται με τεχνητό τρόπο να μην υπάρχουν καθυστερήσεις εκ μέρου των σημερινών φορέων οι οποίοι δεν θέλουν να βελτιωθούν τα πράγματα. Κάτι άλλο σημαντικό είναι η ενιαία πύλη, το one point. Όλοι οι φορείς θεωρούν ότι αυτό είναι αναγκαίο. Η διαδικασία επιλογής προγραμμάτων θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Θα πρέπει να αξιολογούμε τα κόστη και τα πλέον εκτήματα όλων των προτάσεων και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε την εξουσία της Acer στην οποία αντιπροσωπεύονται οι διάφορες εθνικές αρχές. Αυτός ο οργανισμός θα πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και ισορροπημένα τις διάφορες επενδύσεις. Θα πρέπει να λειτουργεί ισότιμα διότι είναι ε, ο μόνος οργανισμός διασφάλισης των συμφερόντων των καταναλωτών θα χρειαστεί να ενισχύσουμε την εξουσία αυτού του οργανισμού Acer, διότι διαφορετικά θα αποδυναμώσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική και θα εκθέσουμε τους καταναλωτές σε αναποτελεσματικές αποφάσεις όπου μόνο μερικά προγράμματα θα βοηθηθούν μόνο σε ορισμένα κράτη-μέλη. Για εμείς, λοιπόν, ε, οι τροπολογίες μας πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, υπάρχει η θέση της Κομισιόν, ε, η γενική θέση της Κομισιόν για τη διαχείριση. Δεν θέλουμε όλα να βρίσκονται στα χέρια μόνο των κρατών μελών, διότι με αυτόν τον τρόπο η διαχείριση γίνεται εθνική. Εμείς ε, επιθυμούμε να υπερασπίσουμε μια ευρωπαϊκή διαχείριση και θα θέλαμε το ίδιο να συμβεί και στο Συμβούλιο. Αλλά σίγουρα πρέπει να υπερασπιστούμε αυτή τη θέση και εμείς στο Κοινοβούλιο. Στην εκθέσή μας θέλουμε επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις περιφέρειες που είναι ενεργειακά απομονωμένες στις απομακρυσμένες περιοχές. Πολλοί μοιράζονται μαζί μας την ίδια ανησυχία. Προτείνουμε λοιπόν μια συγκεντρωμένη πρόταση, όχι ατομική, για κοινά έργα. Βάση ορίων σπουδαιότητας, βαθμίδων σπουδαιότητας ουσιαστικά. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ώστε να μειώσουμε τους προϋπολογισμούς για το Connecting Europe Facility, το μηχανισμό διασύνδεσης της Ευρώπης. Οι ευκαιρίες λοιπόν που θα καθορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προστατευθούν με αυτόν τον τρόπο. Για να ολοκληρώσω ένα ζήτημα για τη χρηματοδότηση. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην δημιουργηθούν διαστρεβλώσεις της αγοράς. Η χρηματοδότηση του Connecting Europe ε, και όσον αφορά ορισμένε υποδομέ που δεν είναι βιώσιμε ε, και που δεν έχουν οικονομικά ωφέλη, αυτέ δεν θα μπορέσουν να επιβιώσει. Σε αυτό λοιπόν το χρηματοδοτικό μέσο θα καταστεί απαραίτητο. Ειδικότερα ε, με τη σημερινή κρίση και ειδικότερα για ορισμένε περιοχέ όπου ο, κίνδυνος, ο πιστοτικό κίνδυνο εμποδίζει την οικοδόμηση υποδομών. Ολοκληρώνω αναφέροντας ότι η πρόταση περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα αλλά εξακολουθεί να εξαρτάται από την καλή θέληση των κρατών μελών για την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να μπορέσει να παρέμβει με μια ενιαία φωνή υπεραμεινόμενο το ευρωπαϊκό όραμα ενισχύοντας την πρόταση που παρουσίασε η Κομισιόν. Θα είμαι φυσικά στη διάθεση των συναδέλφων για μελλοντικές επαφές. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίες. Από όσο καταλαβαίνω από τις τροπολογίες αυτές θα καταφέρουμε να επιτύχουμε πολλά σημεία συμβιβασμού και συμβιβαστικές ψήφους. Ελπίζω λοιπόν ότι κατά τις μελλοντικέ επαφές με του συναδέλφου θα μπορέσω να υπερβώ, να ξεπεράσω τις διαφορές και να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική πρόταση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τον σκιοδησίγητη Ήθελα να σας δώσω πρώτα κάποιες πληροφορίες. Γνωρίζετε ότι υποβλήθηκαν 845 τροπολογίες και ότι συνεπώς ε, έχουμε πολλή δουλειά. Και φυσικά για τις τροπολογίες αυτές θα ακούσουμε πολλές απόψεις. Ε, ξεκινάμε τον κύριο Σαντάργας για την πρώτη παρέμβαση. Ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας, διότι ήδη έχει κάνει πολλή δουλειά. Όπως ανέφερε, πάνω από 800 τροπολογίες ήδη έχουν υποβληθεί στην έκθεσή του όμως έχει προετοιμάσει πολύ καλά τη δουλειά για την επόμενη φάση. Όπως ήδη είπε, Εφόσον ήδη ανέφερε μάλλον ε, τις βασικές κατευθυντήρες γραμμές, τη βασική στρατηγική, ε, εγώ θα ήθελα να εκφράσω κάποιους συλλογισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε την κοινή αγορά. Μιλάμε στο Κοινοβούλιο για την κοινή αγορά και τους μηχανισμούς της. Αλλά την τελευταία δεκαετία κατέστη σαφές ότι σε τόσο σημαντικούς τομείς όπως είναι η ενέργεια δεν μπορεί να λειτουργήσει η ενιαία αγορά χωρίς ενιαία υποδομή. Η κοινή υποδομή είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία της κοινή αγοράς. Στην έκθεσή μας αυτή λοιπόν μας περιμένει ακόμα αρκετή δουλειά όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες. όχι μόνο όσον αφορά την ε, πρακτική διαχείριση της δουλειάς, αλλά για να ε, βελτιώσουμε και την ε, έκθεση. Η βασική δουλειά, λοιπόν, θα γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Καταρχήν, ε, μας ενδιαφέρουν τα έργα κοινού ενδιαφέροντος και οι διαδικασίες επιλογής. Γνωρίζουμε ότι Χρειαζόμαστε συνέχεια τα PCI. Δεν μπορούμε να Δεν μπορούμε να τα επιλέξουμε αυθαίρετα. Θα πρέπει να εξετάσουμε τη σχέση τους με, το, με ένα δεκαετές έργο, για παράδειγμα. Θα πρέπει να δούμε τι αλλαγές μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες. Θα εργαστούμε πολύ πάνω στην σύνθεση των περιφερειακών ομάδων και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι η χρηματοδότηση. Υπάρχει μια παράγραφος στην έκθεση για τη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα εδώ. Είναι πιο ακριβής η παράγραφος, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, μείνουμε σε κατευθυντήρες πάνω στη χρηματοδότηση στην έκθεση αυτή. Αυτά είναι με λίγα λόγια τα βασικά σημεία. Προβλέπω ότι θα πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά ακόμα, αλλά προσβλέπω στην επόμενη φορά που θα έχω την ευκαιρία να συγχαρώ τον εισηγητή, διότι πολλή δουλειά μας περιμένει ακόμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βαλεάν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Κοριέρα Δεκάμπος και κυρία ε, Πρόεδρε. Ε, είχατε δίκιο. Πράγματι μας ε, περιμένει πολλή δουλειά στο θέμα αυτό. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα βασικά σημεία των τροπολογιών μου και ε, τα πολιτικά κίνητρα που με οδήγησαν σε αυτές. Ένα από τα βασικά καθήκοντά μας εδώ είναι να αποφασίσουμε τι προτεραιότητες, σε τι έργα θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε με ε, ευρωπαϊκό χρήμα. Ε, και η έκθεση αυτή σχετίζεται ε, και με τις ε, πολιετής δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Έχω μία τροπολογία για διαγραφή της παραγράφου 15, ακριβώς επειδή πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να αποφασίσουμε δηλαδή τι ακριβώς ε, θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε. Το ε, CEF είναι νέο μέσο και θα πρέπει να ανταγωνιστεί άλλα ε, κοινοτικά προγράμματα και ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πόσα θα λάβει ή αν θα χρηματοδοτηθεί γενικά. Οι κατευθυντήρες γραμμές στόχο είχαν ε, να καθορίσουν ποια έργα θα είναι επιλέξιμα για το καθεστώς PCI. Δεν έχουν να κάνουν με την κατανομή ε, των χρημάτων. Το χρηματοδοτικό μέσο είναι το CF για τον τομέα των μεταφορών. Οι κατευθυντήριες γραμμές ε, σχεδιαγραφούν μια σειρά συγκεκριμένων έργων, ενώ η Κομισιόν ζητά χρηματοδότηση χωρίς να έχει ακόμα σαφή κατάλογο έργων. Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουμε να μην διασφαλίσουμε χρηματοδότηση για την ενέργεια, μην αναφερθώ καν στην τηλεπικοινωνία. Θα πρέπει να έχουμε κατάλογο συγκεκριμένων έργων που σχετίζονται με την ενέργεια ε, και θα πρέπει να είναι έτοιμος μέχρι τα μέσα του 2013. Γι' αυτό Καταλαβαίνω ότι πρέπει να υιοθετήσουμε την έκθεση Κοριέρα όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε αρκετό χρόνο με την έκθεση CEF και να την υιοθετήσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο, ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, άλλες ε, τροπολογίες για την έκθεση αυτή, πέρα από το χρηματοδοτικό θέμα, ε, μπορώ να τα στηρίξω. Ε, ένα από αυτά είναι ο πρώτος κατάλογος των PCI. Επιμένω στην υποχρέωση της ε, Επιτροπής να υποβάλει τον κατάλογο στις περιφερειακές ομάδες για έγκριση, κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου σαφές ε, στο αρχικό κείμενο. Δεύτερον, πιστεύω ότι όλα τα έργα τα οποία είναι επιλέξιμα ως PCI θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις περιφερειακές ομάδες ε, κατά, τη φάση εντοπισμού των προγραμμάτων, ακόμα και αν δεν έχουν ε, συμπεριληφθεί ε, στο σχέδιο του INDP. Επίσης, στις περιφερειακές ομάδες και κατά την ανάπτυξη της μεθοδολογίας TDA θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή. Πιστεύω ότι αυτοί που προωθούν ε, τα έργα έχουν ε, παρκή εμπειρία και ε, αυτό μπορεί να μας προσφέρει μια συμπληρωματική οπτική όσον αφορά το CBA, την ανάλυση κόστους όφελους. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αναπτυχθεί η μεθοδολογία. Σημαντικό πολιτικό θέμα για μένα είναι η διακυβέρνηση στις περιφερειακές ομάδες. Έχω προσπαθήσει να ε, ξεκαθαρίσω κάποιες επιτυχές. Επιμένω ότι οι αποφάσεις ε, για τα έργα PCI θα πρέπει να γίνονται ε, με συνένεση των κρατών μελών ή να μην μπορεί να μπλοκάρει κάποιο κράτος μέλος σε ένα έργο στο οποίο δεν συμμετέχει άμεσα. Ε, επίσης, ε, τα ε, έργα για το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι μια πλήρης εικόνα. 800 τροπολογίες έχουμε. Έχουμε σημαντική δουλειά μπροστά μας. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλές συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο. Το λόγο έχει Σκιώδης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα φυσικά όπως οι συναδελφοί μου να υπογραμμίσω την ποιότητα της εργασίας του εισηγητή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό φυσικά αυτό το κείμενο και βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων που λαμβανούν χώρα στην Επιτροπή αυτή και πρόκειται για μια πρόκληση μεγάλη το να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για αυτό το κείμενο ταυτόχρονα διαβάζοντας τις τροπολογίες που έχουν ήδη υποβληθεί πιστεύω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι ένα κείμενο που αντιπροσωπεύει τις οικολογικές ε, ανησυχίες αλλά πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες θέλουν να αξιοποιήσουν αυτό το κείμενο ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την πορεία μας προς ε, το ευρωπαϊκό οικολογικό όραμα. Υπάρχουν κάποια σημεία ε, στα οποία υπάρχει φιλοδοξία να επιτύχουμε συμβιβασμό. Το πρώτο σημείο είναι ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάλυσης των υποδομών όταν υλοποιούμε υποδομές που θα διαρκέσουν 30, 40, 50 χρόνια. Είναι σημαντικό οι υποδομές αυτές ε, από την κατασκευή τους, ε, από το σχεδιασμό τους να συμφωνούν με τους κλιματικούς ενεργειακούς μας στόχους ε, για το 2050. Το δεύτερο σημείο που υπογραμμίζεται επίσης από αρκετά μέλη αυτής της Επιτροπής είναι η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στον ηλεκτρισμό. Γνωρίζουμε την αξιολογηθήσα αναλογία ε, όσον αφορά τις επενδύσεις, ε, έτσι όπως την έχει αξιολογήσει η Κομισιόν, δύο τρίτα για τον ηλεκτρισμό. Είναι σημαντικό αυτό το κοινοβούλιο να ε, λάβει υπόψη του αυτό το, αυτή την αναλογία δεν μιλάμε εδώ για μια υποδομή μεταφοράς. Ε, θα πρέπει να καλυφθεί από αυτή την έκθεση. Το τρίτο σημείο, επίσης σημαντικό, ε, δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών είναι το ζήτημα των έξυπνων δικτύων και το ζήτημα της διανομής. Καθίσταται σαφές ότι εάν με την ενεργειακή απόδοση και την ευφυΐα των δικτύων αποφύγουμε την κατασκευή ορισμένων υποδομών εξοικονομούμε πολλά και έτσι έχουν αποτέλεσμα οι συζητήσεις που κάνουμε εδώ πέρα στις διαπραγματεύσεις μας ε, όσον αφορά την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Και εκεί θα πρέπει να ενταξούμε το ζήτημα των έξυπνων δικτύων και της διανομής. Τέταρτο σημείο, όσον αφορά τις περιφερειακές ομάδες. Διαφάνεια της εργασίας συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων για εμάς αποτελούν ε, ζωτική σημασία στοιχεία κυρίως για την αποδοχή για το, τον, και για την έγκριση των μεθόδων κόστους και ωφελών και για όλες τις αναλύσεις που θα γίνουν. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν θα ε, οδηγηθούμε σε καθυστερήσεις όλων των προγραμμάτων μόνο και μόνο διότι δεν υπήρξε συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων οι οποίοι θα αμφισβητήσουν τις μεθόδους. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό, το ζήτημα της, ε, του CEF. Και εκεί συμφωνούμε με τη βούληση του εισηγητή να ενισχυθεί η δομή αυτή του μηχανισμού CEF. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια ε, διευρωπαϊκή προοπτική, πραγματική, με ισχυρή εξουσία συντονισμού, ενημέρωσης. Δεν μπορούμε να ε, έχουμε απώλεια απόδοσης ε, λόγω της δομής των υποδομών. Θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματική διευρωπαϊκή δομή συντονισμού. Τελευταίο σημείο όσον αφορά το ζήτημα της αδειοδότησης και της υλοποίησης Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα ζητήματα του περιβάλλοντος, οι κανονισμοί για το περιβάλλον και για άλλη μια φορά θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια, να γίνουν διαβουλεύσεις με τους τοπικούς πληθυσμούς. Ξέρουμε ότι κάθε φορά που ένα πρόγραμμα δεν έχει τη συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών έχουμε ε, τη δημιουργία αντίθεσης σε τοπικό επίπεδο και συχνά ποτέ ε, τα προγράμματα αυτά δεν υλοποιούνται. Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριλάβουμε τους πολίτες από την αρχή στις συζητήσεις αυτές ώστε να αποφύγουμε πολλά προβλήματα. Ευχαριστούμε κύριε Σκεωδησίτη. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Στοζενόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του. Επίσης και από τις τόσες τροπολογίες φαίνεται πόσο δύσκολο είναι το θέμα. Κατά τη γνώμη μου, η ενέργεια θα γίνεται όσο πέραν χρόνος όλο ένα και πιο σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη πολλές φορές στην Επιτροπή μας τα συζητούμε όσον αφορά το τι θα γίνει με τα έργα υποδομής, τι θα γίνει με τα δίκτυα, τι θα γίνει με την παροχή ενέργειας. Βεβαίως και πρέπει να προσέξουμε για το πώς θα μειώσουμε την γραφειοκρατία και θα έχουμε καλύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μια που κάθε έργο στην Ευρώπη προσκρούει στην γραφειοκρατία αυτή. Γίνεται όλο ένα και πιο δυσκίνητη αυτή η διαδικασία. Οπότε γι' αυτό και εγώ έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες. Με αυτές προσπάθησα να βοηθήσω ούτως ώστε η διαδικασία της επιλογής να διακρίνεται από διαφάνεια. Και βέβαια και το να εξασφαλίσουμε το, το πώς θα τηρείται αρχή της υπηκορικότητας. Βεβαίω είναι και εθνική αρμοδιότητα, όπως ορίζουν συνθήκες. Επομένως, τα PCI θα πρέπει να περνάνε από κάποια διαδικασία επιλογής που να διακρίνεται από συνένεση και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να σημειώνεται ομοφωνία και συμμόρφωση μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκομένων περιφερειών. Θα πρέπει επομένω οι διάφορες πολιτικές ομάδες να εξασφαλίσουν μια διαδικασία λήψη αποφάσεων που να διακρίνεται από αποτελεσματικότητα και κάθε τον τρόπο να μην έχουμε πλέον καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων. Θα πρέπει να απλουστευτεί η διαδικασία της επιλογής και όσον αφορά όλα τα στάδια αυτής Έχω υποβάλει λοιπόν σχετικέ τροπολογίε. Είπα θα πρέπει να συντηρηθούν οι διαφορετικέ προθεσμίε που προβλέπονται. Και έτσι πιστεύω ότι οι καθυστερήσεις, οι περιτές θα αποκλειστούν. Επίσης, τα κορυφαία PCI θα πρέπει κατά την προτεραιότητα να ομαδοποιούνται. Θα πρέπει να τους αποδίδεται το ίδιο δικό βάρος γιατί πάρα πολλές φορές είναι δύσκολο κανείς να καθορίζει τις προτεραιότητες όσον αφορά τα σχετικά project γιατί όλα ε, ουσιαστικά έχουν προτεραιότητα και ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση αποσκοπούν οι τροπολογίες μου να προσδεθεί η διαδικασία της επιλογής. να σταματήσουν αυτές οι καθυστερήσεις και επομένως να μην κάνουμε τη διαδικασία ακόμα πιο περίπλοκη και να καθυστερούμε ακόμα περισσότερο από ό,τι σήμερα. Ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώνονται οι ομιλίες των σκιωδών. Ξεκινούν οι ομιλίες των υπολείπων μελών της Επιτροπής. Κυρία Ντεκαστήγιο, Παρακαλώ και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Ντεκάμπρος, τον εισηγητή μας. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, πάρα πολύ αξιόλογο το έργο που επιτέλεσε. Και βλέπουμε το πόσε τροπολογίε έχουν υποβληθεί, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τελικά θα υπάρχει συνένεση γύρω από το κείμενο αυτό. Τώρα να σας πω και εγώ κάτι για τις δικές μας ε, τροπολογίες, αυτές που ε, έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες συναντήσεις. Πρώτον, 108 και 132. Σε αυτές τις τροπολογίες αναφέρεται η συγκρισιμότητα του κόστους, του benchmarking όσον αφορά τις διασυνδέσεις. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Έτσι θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια, έτσι θα προστατευτούν καλύτερα τα συμφέροντα και του κλάδου και των καταναλωτών. Για το 132, για το 129 λέει και πέρα για τα δίκτυα και παράλληλα ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ε, τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιών. Και έτσι να έχουμε μια συνέργεια που θα μας ωφελήσει μεταξύ των δύο ειδών δικτύων. Γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η συνέργεια, αν όχι η πιο σημαντική, το πώς θα αναπτυχθούν εφή δίκτυα ενεργειακά. Τέλος, όσον αφορά τις ε, περιφέρειες, όσον αφορά τους διαδρόμους προτεραιότητας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την τάξη μεγέθους αυτών των έργων, αυτών των προγραμμάτων, το πώς συμμετέχουν. Γι' αυτό και έχουμε την τροπολογία 215. Λέμε εκεί ότι θα πρέπει να πετύχουμε όσο είναι μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, οπότε να μην είναι υποχρεωτικό, να έχουμε περισσότερη ευελιξία, να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χωρίσει αυτές τις περιφερειακές ομάδες και με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε πιο λειτουργικοί, πιο αποτελεσματικοί. Επίσης, Έχουμε την τροπολογία για την χρηματοδότηση που αφορά το άρθρο 15. Η κυρία Βαλιάν μίλησε σχετικά. Και ο κύριος Βάργας, ο σκιώδης ηγέτης του ΕΛΚ, είναι θέμα το οποίο απασχολεί όχι μόνο πολιτικές ομάδες, αλλά και βουλευτές ατομικά. ιδέα εδώ είναι τα κριτήρια της επιλεξιμότητας να εξεταστούν όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές, όσον αφορά την διασύνδεση των ε, ευρωδιευκολύνσεων. Έχει ασχοληθεί με αυτό και η κυρία Γιάλα, όπως ξέρουμε, γιατί μόνο σε αυτά το έργα υποδομής έχουμε μια τέτοια κατάταξη των ε, projects αυτών. Το, το, είπε και η κυρία Βαλεάν. Να δούμε τι θα γίνει με τον κανονισμό για τις συνεργείες υποδομές, για αυτά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος και ε, έτσι να έχουμε ένα ταμείο αλλά θα πρέπει πρώτα πρώτα να ξέρουμε το σχετικό ποσό, αυτό που απαιτείται. Αλλιώ πάμε να διαθέσουμε ένα δισεκατομμύριο χωρίς να ξέρουμε τελικά το πόσο θα χρειάζεται να πρικοδοτηθεί αυτό το ταμείο ε, σύνδεσης ή διασύνδεσης. Άρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το επιχείρημα του πόση θα είναι τελικά η χρηματοδότηση. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία πώς θα κληθούμε να πούμε ποια είναι τα έργα, προγράμματα τα οποία θα χαρακτηριστούν ως κοινού ενδιαφέροντος είτε είναι 9, είτε είναι 5.000, δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί θα πρέπει να έχουμε καθορίσει με, με τρόπο, ε, κάποιο τρόπο τέλο πάντων, τα κριτήρια τη επιλεξιμότητα ανεξάρτητα από το τελικό ποσό τη πρικοδότηση. Γι' αυτό σα λέω. Και υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα, αλλά να μην είμαι Γιατί αν θέλουμε να καθορίσουμε κάποιε προτεραιότητε, κυρία Βαλεάν, κάποια στιγμή αυτό θα το κάνετε όσον αφορά τον οργανισμό. Θα τάξετε κάποιε προτεραιότητε. Αυτό είναι διαφορετικό για τον γενικό κανονισμό. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με έναν κανονισμό ο οποίος θα ισχύει το 2020. Προσοχή, γιατί πρόκειται για ένα θέμα διαρκώ μεταβαλλόμενο και θα πρέπει να διακρίνεται η ρύθμιση από ευελιξία. Άλλο επομένω τα κριτήρια της ε, επιλογή και άλλο το τελικό ποσό. Το ένα δεν πρέπει να επηρεάζει το άλλο. Οπότε δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον σιώδη συγητή του ΕΛΚ και με τον ε, συγητή και με άλλους συναδέλφους σε σχέση με το πόσο, πόσο σωστό είναι να έχουμε τέτοια κριτήρια επιλεξιμότητας για αυτές τις συνεργειακές υποδομές και σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, συναδέλφοι, δεν ήθελα να διακόψω τη συναδέλφο δικαστήριο, αλλά είχαμε ορίσει δύο-τρία λεπτά ομιλίες για τον καθένα και δεδομένου ότι ο κατάλογος των ομιλητών είναι πολύ, μεγάλη, σας παρακαλώ, είναι πολύ μεγάλο, σας παρακαλώ να περιορίσετε το πολύ σε δύο-τρία λεπτά. Τέρεζα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ah, Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη και εγώ να συγχαρώ τον Ντεκάμπος Συμφωνώ με αυτά τα οποία άκουσα σε σχέση με τα βασικά προβλήματα, αυτά που θα πρέπει να επιλύσει η Ευρώπη και να ζητήσει τις λύσεις και συμφωνώ με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι τώρα. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που οποίο το είπαμε προηγουμένως για αυτές τις δύο τροπολογίες που αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι, οι προλαλήσαντες πρώτα-πρώτα να ελευθεί υπόψη το ότι χρειάζεται να έχουμε ε, κάποια υποδιέρεση των ηλεκτρικών διαδρόμων. Επίσης, ε, όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει το κάθε κράτος μέλος για τον κάθε διάδρομο που του αναλογεί και τελικά επομένω να είναι όσο είναι πιο δόκιμη η σχετική κατανομή για να έχουμε την αντιστοίχηση με τα έργα υποδομής. Επίσης, όπως είπε και η κυρία Ντελκαστίγια, να δούμε τι θα γίνει με αυτή την τροπολογία του εισηγητού όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση των χρημάτων που δαπανώνται μια που τώρα περνάμε από αυτή την οικονομική κρίση. Κάτι τέτοιες ώρες είναι δύσκολο κανείς να αποφασίζει σε σχέση με τις δέουσες επενδύσεις. Βεβαίως και όλοι οι και, και όλοι οι καταναλωτές ενδιαφερόμαστε να υπάρχει μια σωστή ρύθμιση και έτσι να εξασφαλιστούν οι πιο καλές υιοθέτηση των πιο σωστών πρακτικών. Και όπως είπε η κυρία Τελικαστήγιο, θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία διάφανη, να προστατεύονται οι καταναλωτέ και να κατοχυρώνονται και τα συμφέροντα του κλάδου. Και είναι πάρα πολύ θετικό το πόσο έχει δεσμευτεί προ αυτήν την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Είναι το λόγο στον κύριο Έλμα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή που κατέστησε πολύ σαφείς τους στόχους αυτού του μέτρου και από όσα λέει καθίσατε πολύ σαφές ότι το κυριότερο κίνητρο είναι το ευρωπαϊκό όραμα και η συγκέντρωση της λήψη αποφάσεων για την ενέργεια και τον έλεγχο της ενέργειας στην Ευρώπη παρά η απόδοση του grid, του δικτύου και η ενεργειακή ε, προμήθεια. Φυσικά όλα αυτά θα γίνουν με τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κράτων μαλλών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να κινείται από τα ίδια τα κράτη-μέλη ε, βάσει του αντιληφθέντος πλέον εκτήματος αυτών των προγραμμάτων και όχι με, από το κέντρο από τις Βρυξέλλες. Λέει ο εισηγητής ότι πρέπει να αποφύγουμε τις διαστρεβλώσεις της αγοράς. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν εκτιμάτε ότι ολόκληρη η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική επιβάλλει διαστρεβλώσεις στην αγορά. Έχουμε αποφασίσει ε, να οδηγήσουμε την αγορά υπέρ της, ε, των καυσίμων χαμηλής ε, εκπομπής ρήπων με αμφίβολες πρακτικές Ακόμη και σε αυτόν τον τομέα έχουμε καθοδηγήσει τις δραστηριότητές μας υπέρ των ανανεώσιμων ενεργειών και κατά της πυρηνικής ενέργειας και δεν βλέπω το λόγο που γίνεται αυτό. Ολόκληρη η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική αφορά τη δημιουργία διαστρεβλώσεων. Συμφωνώ βέβαια με την βούλησή σας να αποφύγουμε τις διαστρεβλώσεις. Ωστόσο αυτή η Επιτροπή και οι πολιτικές της Ευρώπης αφορούν ακριβώς τη δημιουργία διαστρεβλώσεων όσον αφορά το φυσικό αέριο στην Αμερική έχει πέσει στο μισό το κόστος του καθώς ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλύπτουν νέες πηγές φυσικού αερίου και εμείς ε, δεν μπορούμε να το επιδιώξουμε αυτό στην Ευρώπη, δεν τα καταφέρνουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε μείωση τις τιμές του φυσικού αερίου και να εξαρτώμαστε λιγότερο από τις εισαγωγές. Ακούμε ελάχιστα για αυτό το θέμα σε αυτή την εδώ την Επιτροπή. Επίσης σημείωσα μία από τις προτάσεις που εκτίμησα ιδιαίτερα το δικαίωμα των καταναλωτών για αποδοτική και φθηνή ενέργεια. Συμφωνώ μαζί σας, θα ήθελα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε αποδοτική και φθηνή ενέργεια, αλλά αυτό είναι αδύνατο να γίνει με την προώθηση υψηλού κόστους διακοπτόμενων πηγών ενέργειας όπως αιωλική και ηλιακή όπως συνήθω λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως συνήθω συμβαίνει σε αυτή την Επιτροπή και σε αυτό το Κοινοβούλιο εκφράζουμε καταπληκτικές φιλοδοξίες και στη συνέχεια υλοποιούμε πολιτικές οι οποίες καταρρύπτουν αυτές τις φιλοδοξίες και τις καθιστούν μη επιτεύξιμες. Είμαι λοιπόν αντίθετος με αυτό το ε, μέτρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο συνάδελφος Γκίρεκ, παρακαλώ. Γκίρεκ, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, μα μας μπερδεύουν πάντα με τον συναδέλφο Γκίρεκ. Ε, ίσως να έχετε εσείς το λόγο, ε, ζητώ συγγνώμη. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Του εύχομαι καλοκουράγιο για ε, τη μελέτη των 800 και τροπολογιών και εγώ συνεισέφερα. Θα ήθελα να επισημάνω τρία προβλήματα. Πρώτα απ' όλα το θέμα των περιφερειακών ομάδων. Ο κύριος Κιώδης και οι υπόλοιποι έχουν δίκιο όταν λένε ότι οι δραστηριότητες αυτών των περιφερειακών ομάδων θα πρέπει να, είναι, να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Όσον αφορά τις δικές μου τροπολογίες, θεωρώ ότι δεν πρέπει να παρεμποδίζονται οι δραστηριότητες αυτών των ομάδων ώστε να μπορούν να κάνουν προτάσεις επενδυτικές προς την Κομισιόν για την υλοποίηση μελλοντικών έργων. Μια δεύτερη ομάδα τροπολογιών αφορά την αντικειμενικότητα όσον αφορά τις μεθόδους επιλογής θα πρέπει να υπάρχει επαρκής πίνακας αξιολόγησης ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των προγραμμάτων. Φυσικά πρέπει να δούμε και τη σχεση κόστου κόστους-οφέλους όσον αφορά την επιλογή έργων διότι σε αυτή τη βάση τα κράτη-μέλη ε, καθορίζουν τις τα ενδιαφέροντα προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε αυτά τα προγράμματα από άποψη εκτέλεσης. Τρίτον, όσον αφορά την αξιολόγηση εξ αυτών των έργων των υστέρων αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων, πραγματοποιούμε αναλύσει, απόδοσης, κόστου ωφέλου εκ των προτέρων. Αλλά πιστεύω ότι οι επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει θα πρέπει επίσης να αξιολογούνται ώστε να ε, διαπιστώνουμε τις επιπτώσεις για τις αγορές. Πρέπει να βλέπουμε τις συνολικές επιπτώσεις των και συνέπειες των επενδύσεων. Καλό λοιπόν τον κύριο Σιγητή να λάβει υπόψη του τις τροπολογίες μου και το ευχόμαι με καλή επιτυχία. Ευχαριστώ κύριος άντρας, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ο οργανισμό, τόσο ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε του στόχου εκείνου που ανέκαθεν είχαμε τάξει και που δεν καταφέραμε ακόμα να υλοποιήσουμε. Να υπάρχει δηλαδή μια εσωτερική μια ενεργειακή αγορά. Δυστυχώ. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε αυτό τον στόχο τον οποίο έταξε το Συμβούλιο το 2002 και ανανέωσε την υποχρέωση το 2010 ε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κατάλληλη παραγωγή ενεργείας για πλευράς μελλον. μελών. Γι' αυτό θα πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε την όθηση που πρέπει στα έργα υποδομής και κυρίως στο θέμα των διασυνδέσεων. Πάρα πολύ αξιολογή αυτή η έκθεση, όπως όλοι είπαμε και δεν θα ξέρει τι να κάνει με τόσο τόσο συγχαρητήρια ο κύριος Κάμπος. Όλα αυτά τα συγχαρητήρια πάντως τα αξίζει. Έχουμε μια, ένα σωρό αξιόλογες τροπολογίες, τόσο ώστε να επιφέρουμε βελτιώσεις σε αυτό το αξιόλογο κείμενο και αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ε, οι διατάξεις οι με την αποθήκευση ενεργείας. Και τι θα γίνει επίσης με την μεταφορά της ε, ενεργείας δεδομένων της, ε, της οργάνωσης της αγοράς των, των φορέων που μεταφέρουν ενέργεια. Άρα τελικά θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ε, απάνες που αναδύονται. Διότι στο παρελθόν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και αν το κόστος αυτό είναι πολύ πάνω του φυσιολογικού, τότε θα πρέπει αυτός που θα έχει αναλάβει το έργο να παράσχει τι κατάλληλε εξηγήσει. Πάντω είναι ξεκάθαρο ότι Εάν η εκτέλεση του έργου καθυστερήσει, τότε ο εργολάβος θα πρέπει να φέρει την ευθύνη ανάλογα με το εάν εκείνος ευθύνεται για την ε, καθυστέρηση ε, και η καθυστέρηση οφείλεται στην κακή διαχείριση του για να είμαστε άδικοι. Άρα θα πρέπει να δούμε με τι ρύθμιση θα αποφύγουμε δυστρεβλώ στην αγορά, γιατί θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει μόνο τα έργα κοινού ενδιαφέροντος ε, τα οποία από πλευράς κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής πρόκειται να, ε, να ωφελήσουν ε, με τρόπο που δεν θα μπορούσαμε να ωφεληθούμε με άλλο τρόπο. Πάντως, προς τον κύριο Χέλμερ και στον κύριο Ζαντό, έχω να πω τα εξής με, με, κάθε, με κάθε συμπάθεια προς τις θέσεις τους και πάρα πολύ φιλικά έχω να τους πω ότι εν μέρει έχουν δίκιο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούν οι συνάδελφοι ότι πάρα πολλέ από τι πολιτικές τους ώστε που αποσκοπούν στην μείωση του, του, άνθρακα ε, θα πρέπει να είναι συμβατές με την αναγκαιότητα του να είμαστε ανταγωνιστικοί και θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει και την σωστή ε, παροχή ενέργειας. Και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνούμε για να είμαστε σωστοί. Για τον κύριο Ζαντό τώρα, στα γαλλικά, φίλε Ζαντό, έχω να σου πω το εξή. Τόνισε το ότι θα πρέπει η ηλεκτρική ενέργεια να αποτελεί μία προτεραιότητα. Σωστό. Να μην ξεχνούμε όμως ότι αν έχουμε ένα ενεργειακό σύστημα όπου θα χρησιμοποιούνται πάρα πολύ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την συνέχεια, μην έχουμε ε, διακοπές στην υπαρχία της ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο. Και εκεί υπάρχει συμπληρωματικότητα όσον αφορά τα έργα υποδομής. Να μην τα ξεχνούμε αυτά. Αλλιώς τότε δεν έχουμε την συνολική εικόνα του τοπίου. Κάτι άλλο επίσης. Κάντε μου μια χάρη. Αναφερθήκατε στις δυσκολίες και, τα εμπόδια που βάζουν τα τοπικά σημεία καθώς στην εκτέλεση των, έργων. Όμως, οι ομοειδεάτες σας προκαλούν αυτά τα προβλήματα. Εσείς τους ξεσηκώνετε. Τουλάχιστον στην Ισπανία, οπότε παρακαλώ, στη χώρα μου πηγαίνετε και πείτε στον κόσμο ότι αυτά τα έργα υποδομής χρειάζονται, είναι πολύ σημαντικά για όλη την Ευρώπη και ότι πρόκειται όλους να μας ωφελήσουν. Αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και στον πρωτό σας ευχαριστώ που θα τους το πείτε. Ευχαριστώ. Ζήτησε το λόγο η κυρία αλλά δεν τη βλέπω η κυρία Κουράσκα που e, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα φυσικά να συγχαρώ τον εισηγητή Ταυτόχρονα θα ήθελα να του ζητήσω να λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις που προετοίμασε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. στο θέμα που συζητάμε σήμερα σχετίζεται στενά με την περιφερειακή πολιτική, με τα περιφερειακά ταμεία, με τα ταμεία που θα επηρεαστούν από κάποιους ε, στόχους ε, και μία σειρά απολύσεις και αποφάσεις που θα υποχρεωθούν να λάβουν ε, η Περιφερειακή Φορήση η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη συζήτηση και εγώ ίδια συμμετείχα σε αυτή τη συζήτηση, υπέβαλα πολλές τροπολογίες. Θα σας ζητήσω λοιπόν να τις λάβετε υπόψη σε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας εκείνης. Εκφράστηκαν πολλές ανησυχίες όσον αφορά το μέγεθος αυτών των προγραμμάτων προγράμματα στα οποία συμμετέχουν πολυάριθμα κράτη-μέλη και όπου η διαχείριση των ε, προγραμμάτων αυτών είναι ουσιαστικά αδύνατη. Κατά την άποψή μας θα πρέπει να προσανατολιστούμε σε πιο μικρά προγράμματα, μικρότερου μεγέθους. Αυτό είναι από τα συμπεράσματα, τα δικά μου. Δεν ε, έχει γυρίσει η κυρία ναι δεν έχει γυρίσει. Το λόγο έχει ο κύριο εισηγητής ε, και σα συγχαίρω και εγώ ε, μαζί με όλα τα συγχαρητήρια που δεχθήκατε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ίσως θα έπρεπε να σας πω τι γίνεται με τα ηλεκτρικά οχήματα. Δεν ξέρω αν εξαιτίας αυτών έλαβα τόσους επένους. Ε, είναι πάντως ε, ένα θέμα το οποίο έχει δεχτεί και επικρίσεις ε, και επένους. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τις παρεμβάσεις τους, ιδιαίτερα τους σκιώδεις εισηγητές διότι αυτοί είχαν περισσότερο χρόνο να εξετάσουν ε, αναλυτικά την έκθεση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που, έχει, που έχετε δείξει για το θέμα αυτό. Θα πρέπει, όπως είπανε πολλοί, να γίνουν ε, σημαντικές επενδύσεις ε, σε, υποδομής, ε, σε υποδομές και μάλιστα μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να το σχεδιάσουμε αυτό πολύ προσεκτικά. Προς τον συνάδελφο Ζαοτάκας να πω ότι είμαι ευγνώμων που μπορεί να συμφωνήσει με πολλά από τα θέματα που έχω παρουσιάσει. Όσον αφορά τις περιφερειακές ομάδες, ε, τις οποίες ε, ανέφεραν και, και οι τελευταίοι ομιλητές, η κυρία Τεκαστήλιο και άλλοι, ε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει τονιστεί. Το θέμα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία να την απλοποιήσουμε. Ε, ίσως να μην συμμετέχουν όλες οι χώρες, ε, να λειτουργούμε σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να διατηρούμε την ευρωπαϊκή οπτική. Μπορώ να συμφωνήσω και με τον συνάδελφο Σαουτάκας όσον αφορά την χρηματοδότηση και τις ε, γενικές κατευθυντήρες γραμμές προς τη συνάδελφο Βάλεαν. Να την ευχαριστήσω για την υποστήριξή της όσον αφορά τον ε, πρώτο κατάλογο αυτών των PCI, των ε, έργων κοινού ενδιαφέροντος. Ε, αναφέρεται στην ανάλυση κόστους, ωφέλους και τις περιφερειακές ομάδες. δεν μπορώ να συμφωνήσω με όλες τις, τις θέσεις. καταλαβαίνω την επιχειρηματολογία της στο θέμα αυτό. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν ενδεχομένως ε, τον ε, Σεπτέμβριο να εξετάσουμε τριμερό το θέμα αυτό. Κάτι με το οποίο δεν μπορώ να συμφωνήσω ιδιαίτερα από αυτά που είπε η κυρία Βάλεαν είναι η διαγραφή του άρθρου 15. Εάν ε, το να αφαιρεθεί δηλαδή το εδάφιο από, το, συγκεκριμένο τη νομική πράξη και να υπάρχει μόνο, στο, μέσω ε, μόνο στη διευκόνηση CEF, το συνδέοντας στην Ευρώπη. εάν ε, αφαιρέσουμε τους βασικότερους στόχους ε, από την έκθεση αυτή, τότε δεν έχει νόημα η όλη εκπονησή της. Και μας ενδιαφέρει και η όλη λογική της διευκόλυνσης συνδέοντας ε, την Ευρώπη. Μας ενδιαφέρει επίσης η αιτιολόγηση ε, κατά την ε, διαδικασία επιλογής αυτή τη στιγμή. δεν διαφωνώ με αυτά που λέτε για το άρθρο 15, αλλά μπορούμε να το ε, επαναλαμβάνουμε σε διάφορες νομικές, νομικές πράξεις. Ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με κάτι τέτοιο. Εάν όμως αφαιρέσουμε τελείως ε, την παράγραφο αυτή, το άρθρο αυτό από την νομική πράξη αυτή, αυτό δεν θα αποτελεί βελτίωση του κειμένου. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Ζαντό για τις παρατηρήσεις του. Δεν πρόκειται για οικολογικό κείμενο, πηγαίνει όμως προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω μαζί του και όσον αφορά τις προτεραιότητες για το ηλεκτρικό ρεύμα. Εάν θέλουμε να υποστηρίξουμε την ηλεκτροδότηση, θα πρέπει να μιλάμε και για άλλα πράγματα εκτός από την αποδοτικότητα της ενέργειας. Θα πρέπει να μιλάμε και για ε, λιγότερο διπένουσες ε, πηγές θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις στον τομέα της ενέργειας. Καθότι έχουμε ακόμα σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την αποθήκευση μέσα στα δίκτυα. Μπορώ να συμφωνήσω και με τις προτάσεις για τα smart grids, τα FEE δίκτυα, καθώς και όσον αφορά την διαφάνεια των περιφερειακών ομάδων. η έννοια της διαφάνειας και η συμμετοχή των ε, περιφερειακών και εθνικών φορέων είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και εμάς. Θα μας απασχολήσει και όταν ασχοληθούμε ε, στο μέλλον με προβλήματα. Υπάρχουν ε, διάφορες εναλλακτικέ λύσεις. Μέρος των υποδομών θα μπορούσε να κατασκευαστεί υπογείως, κάτι το οποίο είναι το οποίο στοιχίζει πιο πολύ, ο συνάδελφος Κοζενόφσκι ανέφερε δύο σημαντικά θέματα. Μπορώ να συμφωνήσω με το πρώτο, ότι θα πρέπει ε, να απλοποιήσουμε όσο μπορούμε τις ε, διαδικασίες, ενώ με την ε, δεύτερη του παρατήρηση δεν μπορώ να συμφωνήσω τόσο πολύ όσον αφορά τις προτεραιότητες και την ισορροπία. Φυσικά θα πρέπει να κάνουμε τις αναλύσεις κόστους όφελους. Θα πρέπει να εξετάζουμε την αποδοτικότητα. Δεν είναι δυνατόν να ε, τα δούμε όλα με την ίδια οπτική. Ε, ευχαριστώ την ε, κυρία Τερκαστήγιο για τις πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις της. Είπατε ότι μακρηγορήσατε, αλλά για μένα ήταν χρήσιμα αυτά που είπατε. Και μπορώ να συμφωνήσω με τις ε, συστάσεις σας όσον αφορά τις ομάδες προτεραιοτήτων. Ε, και συμφωνείτε εσείς με τη διατήρηση του άρθρου 15. Άλλο θέμα είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας το οποίο αποτελεί ένα μέρος ε, των αρμοδιοτήτων ε, του Κοινοβουλίου. Στο Κοινοβούλιο δεν ασχολούμαστε με το ίδιο το προϊόν, ούτε με τις ε, λεπτομέρειες του προϊόντος. Ασχολούμαστε με, τις, με τους κανόνες. Μας ενδιαφέρει οι γενικές αρχές να είναι καλές. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας αυτές. Σας ευχαριστώ και για την υποστήριξή σας. μπορώ να συμφωνήσω με τις ιδέες σας και να σας ευχαριστήσω και την υποστήριξη όσον αφορά τη διαφάνεια των δαπανών και όσον αφορά το benchmarking. Επίσης, ε, ήταν πολύ χρήσιμη η ε, παρέμβαση του συναδελφού Ντεμέγερ δεν συμφωνώ απόλυτα ότι ε, η ευρωπαϊκή στρατηγική ε, αποδυναμώνεται. Ούτε το θέμα είναι να τα, να όλα οι Βρυξέλλες. Το θέμα είναι ότι θέλουμε αποδοτικότητα. Θέλουμε καλά αποτελέσματα και η ευρωπαϊκή πολιτική δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά. Μεγαλύτερες στρεβλώσεις στην αγορά θα έχουμε αν δεν έχουμε ενιαίες δαπάνες ε, για την ενέργεια. Και διαπιστώθηκε στις Ηνωμένε Πολιτείες πόσο σημαντικό είναι το φυσικό αέριο. Και μπορεί κανείς ε, να παράγει ε, ε, με κόστος 2 δολάρια την μονάδα, ενώ στις, στη Ιαπωνία το κόστος είναι 17 δολάρια. Υπάρχει το θέμα τη, του αερίου από σχιστόλιθο, αλλά κανείς δεν γνωρίζει πόσο μεγάλα είναι τα αποθέματα. Ε, και γενικά τα αποθέματα μειώνονται σημαντικά. Ε, δυστυχώς δεν σημείωσα το όνομα του επόμενου συναδέρφου, ο οποίος ε, συμφώνησε με τις παρατηρήσεις για τις περιφερειακές ομάδες. Αναφερθήκε και στον εκ των υστέρων έλεγχο. Ε, αυτό είναι κάτι χρήσιμο για τα έργα τα οποία θα πραγματοποιηθούν. μπορεί να θεωρεί... Επίσης, μια παρατήρηση, Λίδα Κουάτρα, ε, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και θα ήθελα ε, τέλος ε, να φτάσω στις παρατηρήσεις του συναδέρφου Πρόβνικ. Μεταξύ περνάει ο χρόνος, θα σα ζητήσω να είστε πολύ σύντομο. Ναι, ουσιαστικά έχω πει τα... όλα όσα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους. Ευχαριστούμε πολύ για τις ε, πολύ ολοκληρωμένες απαντήσεις, τις παρατηρήσεις που ακούσαμε. Ο πρόσωπος της Κομισιόν, κύριε Βενουά, σας παρακαλώ να είστε εξαιρετικά σύντομος, διότι ε, προσπαθούμε να συζητήσουμε πολλά θέματα σήμερα. Θα έχετε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσετε αυτή τη γνωμοδότηση πιο εκτεταμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα φυσικά να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του και για όλο, το έργο όλων των μελών αυτής της Επιτροπής. Όλοι μαζί, εκτός από τον κύριο Έλμερ φυσικό, συμμεριζόμαστε τους στόχους και κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να περιοριστώ λοιπόν σε ελάχιστα σχόλια Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την αναγνώριση των PCI, των προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος, αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι ποια έργα θα χαρακτηριστούν ως κοινού ενδιαφέροντος. Έχουμε συμφωνήσει ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι διαφανής. Αλλά έχουμε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τη σύνθεση των περιφερειακών ομάδων θα πρέπει να έχουν σαφή καθήκοντα και να έχουν ε, λειτουργικό μέγεθος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόντων ε, στο έργο άμεσα είναι αδύνατο από πρακτική άποψη και αυτό σχετίζεται με τις τροπολογίες 702, 703, 708 και 713. Αλλά φυσικά η διαφάνεια θα πρέπει να διασφαλίζεται και πιστεύουμε ότι ανοιχτές διαβουλεύσεις και η δημοσίευση των πληροφοριών όπως ε, ε, ζητάνε οι τροπολογίες 725 έως 728 είναι σωστή προσέγγιση. Όσον αφορά την υλοποίηση των έργων κοινού ενδιαφέροντο, είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο θέλει να δει την έργα αυτά ολοκληρωμένα και θα πρέπει να φροντίσουμε να διασφαλιστεί αυτό. Αυτό μπορεί να έχετε πιθανώς σε διένεξη με το Συμβούλιο όπου θα ήθελαν να μην υπάρχουν περιορισμοί διασφάλισης της υλοποίησης των προγραμμάτων όσον αφορά την αδειοδότηση. Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει μια επιταχυμένη διαδικασία διότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη υλοποίησης αυτών των υποδομών. Ε, υποστηρίζουμε πολλές από τις τροπολογίες αλλά θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία να διατηρηθούν οι προθεσμίες ε, όπως ορίζονται και η έννοια του one-stop shop. Είναι σαφές ότι όλα αυτά και σχετίζονται και με την καλύτερη διαφάνεια και καλύτερη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων πληθυσμών. Πιστεύω ότι και σε αυτό το σημείο εμείς ε, συμμεριζόμαστε με την ανησυχία των πρασίνων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες ε, στις αρχές ενός προγράμματος κατά το σχεδιασμό του και ότι αυτό θα επιτρέψει ε, τη συντόμευση της διαδικασίας αδειοδότησης τώρα όσον αφορά τη χρηματοδότηση το γνωστό άρθρο 15 υποστηρίζουμε τη θέση του εισηγητού είμαστε κατά τη διαγραφής του άρθρου 15 Θέλαμε επίσης να πούμε στην κυρία Βαλέαν ότι αυτή η συζήτηση έχει λάβει χώρα ήδη στο Συμβουλίο και έχουμε πείσει τα κράτη-μέλη ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές για, τη διευρωπαϊκά ενεργειακά, για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές είναι μια ολιστική προσέγγιση που καλύπτει τέσσερα στοιχεία τα οποία πρέπει να διατηρούνται μαζί. Δηλαδή αναγνώριση των προτεραιοτήτων, αδειοδότηση, η διαδικασία κατανομής επιμερισμού του κόστους που πρέπει να γίνεται πριν από οποιαδήποτε χρηματοδότηση με χρήματα των φορολογουμένων. Και εκεί τίθεται το ερώτημα. Το ζήτημα το ότι πρέπει αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές να διατηρούνται συνεκτικές. Γι' αυτό το άρθρο 15 θα πρέπει να υπάρξει σε σχέση με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές που σχετίζονται με τη διαδικασία καταμερισμού του κόστους. Επίσης, είμαστε αντίθετοι οποιασδήποτε εκ των προτέρων εκχώρησης κονδυλίων θα πρέπει να διατηρήσουμε τη μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ των τομέων όπως εμπορική βιωσιμότητα, ανάγκη χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι άμεσα αναλογική ανάλογη με τις ενεργειακές ανάγκες. Ο ενεργειακός τομέας είναι διαφορετικός από τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες. Και εκεί φυσικά η παρούσα Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ιδιαιτερότητες οι ενεργειακές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Συμφωνώ επίσης ότι η υλοποίηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου αποτελεί σημείο Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, είμαστε κατά της ε, χρηματικής υποστήριξης για υποδομές ε, ε, πετρελαϊκές. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιοριστούμε σε προγράμματα Smart Grid διευρωπαϊκά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Προβλέπεται ψηφοφορία στις 19 Ιουνίου, όπως γνωρίζετε. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Σας υπενθυμίζω ότι θα βρείτε στο υλικό και τα πρακτικά του workshop που έλαβε χώρα τέλη Μαρτίου. Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση για τον ενεργειακό χάρτη πορείας για το 2050. Το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Τζαβέλα που είναι η συγγήτρια και στη συνέχεια οι υπόλοιποι έχουμε προβλέψει περίπου 50 με 60 λεπτά. σε, παρακαλώ λοιπόν να λάβετε την ευθύνη για τον περιορισμό των ομιλιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ο δικός χάρτης ενέργειας 2050 Είναι θέμα ιδιαίτερα σημαντικό. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Το πρόβλημα είναι ότι όσοι μιλάνε δεν ακούνε. Είναι θέμα ιδιαίτερη ε, σημασία δεδομένη ε, τη ε, μακροπρόθεσμη προοπτική του και δεδομένης της, της ε, συγκεκριμένης χρονικής στιγμής η ενέργεια η ενέργεια παίζει πολύ συγκεκριμένο ρόλο και για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θέλω να τονίσω ότι βλέπουμε το θέμα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Μας ενδιαφέρει η βιομηχανία, η έρευνα και η ενέργεια. Σημείο 1. Πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ανταγωνιστικές ε, τις ε, βιομηχανίε μας στον τομέα της ενέργειας. Δεύτερον, πώς μπορούμε να πετύχουμε ε, ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση. Και τρίτον, ποιες είναι οι μελλοντικέ τεχνολογίες που θα χρειαστούμε για να πετύχουμε τους στόχους μας και ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες μας στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Έχει τονιστεί το θέμα ε, της ε, μείωσης των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα, ιδιαίτερα από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Θέλουν να πετύχουν μείωση σε ποσοστό 80 με 90% μέχρι το 2050 από τις βιομηχανοποιημένες χώρες ως ομάδα. Αυτή είναι πολύ μεγάλη πρόκληση δεδομένων των, διαφορο... των διαφόρων χαρακτηριστικών των των ενεργειακών τομέων των χωρών αυτών. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε το όφελος προς ε, τα κράτη-μέλη ε, της ε, συνεργασίας με στόχο μεταρρύθμιση των ενεργειακών συστημάτων τους. Αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα και αυτόν τον χάρτη πορείας για το 2050 θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως βάση για να προτείνουμε πρωτοβουλίες ε, στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής ε, με στόχο την ε, πρόταση ενεργειακής πολιτικής για το 2030 με συγκεκριμένους στόχους. Αναγνωρίζω ότι μεταξύ των ευρημάτων του ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050 υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία σε διάφορα σενάρια τα οποία θα, θα είναι απαραίτητα για την μεταρρύθμιση του ενεργειακού συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης άσχετα από το ξεχωριστό δρόμο που θα επιλεγεί για να πετύχουμε ένα ε, σύστημα ε, με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πιστεύω λοιπόν ότι η αποδοτικότητα της ενέργειας ε, και η υποδομή της ενέργειας αποτελούν θέματα στα οποία δεν μπορούμε να μετανιώσουμε. Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα ήθελα να τονίσω ότι μια πιο ολοκληρωμένη ε, ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας είναι απαραίτητη. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν ώστε να βελτιστοποιήσουν ε, το, την αναλογία κοστου όφελου ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να φροντίσουμε να γίνονται επενδύσει εκεί που θα είναι πιο παραγωγικέ και αποτελεσματικέ. Ε, ενώ τα κράτη-μέλη ε, επιδιώκουν τον στόχο της ανεξαρτησίας ε, της ενέργειας, θα πρέπει να επιδιώξουμε και τον στόχο της εξάρτησης μεταξύ μας, δημιουργώντας grids, δίκτυα δηλαδή, τα οποία να συνδέονται το βορρά με τον νότο και την ανατολή με τη δύση. Ε, εγώ προέρχομαι από νότιο κράτος μέλος ε, και με ανησυχεί ιδιαίτερα ε, με ανησυχούν ιδιαίτερα, με απασχολούν ιδιαίτερα οι εξελίξεις στον νότιο διάδρομο. Τέλος, το 2050 θα αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις και θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωση της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2014. Γιατί, διότι κοιτώντα και τους δικούς μας πόρους, όταν μιλάμε για ενεργειακή διαφοροποίηση ε, και, με, ε, και την ενεργειακή ασφάλεια, υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ευέλικτους πόρους ε, στο σύστημα ενέργειας και υπάρχει ανάγκη ε, να έχουμε επαρκή, ε, ε, επαρκές δυναμικό ώστε να διασφαλίσουμε την, την παροχή ενέργειας. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και το φυσικό αέριο διότι και τα δύο αυτά είναι σημαντικά για το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης. Κυρία Πρόεδρε, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Πιο πολύ με ενδιαφέρει να ακούσω τι έχουν να πούν οι άλλοι μου συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ εσάς. Ξεκινάμε τον κατάλογο των σκιωδών. Θα μπορούσα να σας δώσω τρία λεπτά, αν συμφωνείτε. Ε, ρυθμίστε το όπως θέλετε εσείς, κύριε Ρόη, παρακαλώ. Äh, Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια, ευχαριστώ και την Επιτροπή. Πιστεύω ότι είναι πολύτιμο το εγγραφό της, διότι για πρώτη φορά δεν ε, επιλέγουμε έναν πολιτικό δρόμο, αλλά ε, παρουσιάζονται διάφορα σενάρια και έτσι ε, γίνεται σαφές ότι με το βλέμμα στο 2050 που δεν γνωρίζει κανείς τι θα συμβεί μέχρι τότε, έχει τη δυνατότητα κανείς να αξιολογήσει τις ε, διάφορες ε, πιθανές εξελίξεις. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα σας παρακαλούσα την ε, διαφάνεια, την αντικειμενικότητα του εγγράφου αυτού να μην την αραιώσουμε, να μην την αποδυναμώσουμε προσπαθώντας να κάνουμε τους έξυπνους. Ε, η Κομισιόν ε, τονίζει ότι ε, στην, όσον αφορά την απόδοση της ενέργειας υπάρχει, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες. Όχι εξοικονόμηση, αλλά απόδοση. Σημαντικό είναι να συνειδητοποιούμε ότι είναι θέμα μεθόδου. Πιο καλό θα είναι να ε, ε, να εκμεταλλευτούμε ε, αυτό που είναι η δύναμή μας στην Ευρώπη, η ηγετική μας θέση στην τεχνολογία. Αυτό είναι το θετικό της Ευρώπης, όχι οι οικονομίες που υπαγορεύουν τους ίδιους κανόνες για όλους. Επίσης, χρειαζόμαστε μία ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ε, τα ε, εθνικά συστήματα ε, προώθησης ουσιαστικά σπαταλούν χρήματα. Εάν χρειαζόμαστε ένα μεγάλο έργο με χαμηλό κόστος και μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον, πρέπει να το κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν γίνεται αποτελεσματικό αυτό σε εθνικό επίπεδο. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να να, να αλλάξουμε και να πούμε ότι θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε κάτι τώρα. Και τρίτη μου παρατήρηση, συμφωνώ ε, με την Κομισιόν που λέει ότι δεν θα, δεν θα πετύχουμε τους στόχους αυτούς εάν ποντάρουμε μόνο σε ένα είδος ενέργειας. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Αυτό είναι απόλυτα σωστό από κράτος μέλος σε κράτος μέλος ε, θα δοθεί ε, διαφορετική απάντηση στο θέμα αυτό. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας δρόμος, ε, όχι, δεν είναι τα πάντα όμως και ο άνθρακας μπορεί να παίξει ρόλο στο μέλλον κατά την παροχή ενέργειας και όσον αφορά την ε, δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα και εδώ θα πρέπει ε, τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα ε, να θεσπίσουν ανάλογους νόμους και ξέρω γιατί πράγμα μιλάω διότι το δικό μου κράτος μέλος κάνει σημαντικά λάθη στον τομέα αυτών και όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια δεν χρειάζεται να την αγαπήσει κανείς αλλά αν θέλει κανείς πολλή ενέργεια χωρίς ε, επιπτώσεις στο, στο περιβάλλον κλπ. Ε, δεν θα καταφέρουμε να παρακάμψουμε την πυρηνική ενέργεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Ρόιλ. Το λόγο έχει η συνάδελφος Βαν Μπρέμ της Κιώδης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ επίσης, κυρία Τζαβέλα, για την παρουσίαση. Σίγουρα η συζήτηση θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας ε, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Συμφωνώ με τον συναδέλφο Ροέλ ότι η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και η μελέτη της θα είναι ενδιαφέρουσα. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η Επιτροπή θα μπορέσει να καταλήξει σε συμπέρασμα ώστε να επιτευχθεί το όρομα για το 2020, 30 και 50. Πρόκειται για ένα καθήκον ε, δικό μας στο Κοινοβούλιο, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να καθορίσουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους. Σίγουρα η Κομισιόν ε, μας έδωσε να καταλάβουμε ότι στο ενεργειακό σύστημα χρειάζεται να υπάρχει μια εγγύηση εφοδιασμού και μετά μέχρι το 2050 θα χρειαστεί να ε, προσθεθούν συγκεκριμένα ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, και μείωση κατά 95% των ε, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Όλα αυτά θα γίνουν σε συνδυασμό με μια ανταγωνιστική οικονομία μέχρι το 2050. Αν αυτός είναι ο στόχος τότε γνωρίζουμε ακριβώς ποιο είναι το σενάριο που προτείνει η Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε για αυτό το σενάριο, αλλά πρώτα απ' όλα αυτό το σενάριο πρέπει να είναι βιώσιμο. Ήθελα να υπογραμμίσω, όπως και στην προηγούμενη συζήτηση, ότι οι υπάρχουσε αυτή τη στιγμή υποδομές είναι παλιές. Αυτό είναι θεμελιώδη σημασίας, διότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να λάβουμε αποφάσεις. Όσον αφορά τους στόχους 2020 θα πρέπει να τους επιτύχουμε και θα πρέπει ίσως να τους ενημερώσουμε. Πρέπει να συζητήσουμε και να καθορίσουμε για τους στόχους επίσης του 2030 για τον ενεργειακό τομέα. Τι θα πρέπει να είναι δεσμευτικό για τα κράτη-μέλη, διότι όπως γνωρίζουμε όλοι η ενεργειακή απόδοση αποτελεί πάντα θέμα συζήτησης σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Φυσικά όμως θα πρέπει να καταλήξουμε και σε μια καλή συμφωνία με το Συμβούλιο για αυτό το τομέα, κύριος, για τους μακροπρόθεσμους στόχους. Ο συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης ε, θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για μας. Τρίτη αρχή που θα ήθελα να υπογραμμίσω και που μου φαίνεται σημαντική, όπως έχει ήδη εποθεί στην Ευρώπη, υπάρχει μια σειρά από υποδομές, είτε μιλάμε για πυρηνικές, ε, είτε στον τομέα του άνθρακα ή του φυσικού αερίου, αλλά θα πρέπει να ληφθούν νέε αποφάσεις. Αποφάσεις που θα χρειαστούν 20, 30, 40 χρόνια και όλες αυτές θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους μας για το 2050. Ε, σίγουρα πρέπει να καθορίσουμε σαφώς την περίοδο μετάβασης, έχοντας υπόψη μας επίσης τα καύσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο μεταξύ, στο ενδιάμεσο ώστε να υπάρξει μια σωστή μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο φυσικό αέριο και ούτω καθεξής. Φυσικά πρέπει να πω ότι όπως φαίνεται υπήρξε ένα άρθρο ιδιαίτερα ενδιαφέρον όπου αναφερόταν ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο για παράδειγμα είχαμε πολύ αέρα, πολύ ήλιο και είδαμε ότι καταναλώθηκε πολύ λιγότερη ενέργεια άλλης φύσης. Τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι σημαντικό να έχουμε, για παράδειγμα, ε, κατάλληλους σταθμούς παραγωγής ε, ε, για παράδειγμα φυσικού αερίου που θα μας επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση προς τους στόχους μακροπρόθεσμα. Επίσης πρέπει να προβούμε σε ανάλυση κόστους ωφελών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των διαφορών μορφών ενέργειας ε, που θα χρησιμοποιούμε σκεπτόμενοι τις πρώτες και μετά την οικοδόμηση των κέντρων παραγωγής και την παραγωγή της ενέργειας. Τέλος, αντιλαμβάνομαι ότι μακρηγόρησα λίγο, θα προσπαθήσω να το πω εν συντομία. Ήθελα να μιλήσω και για το ε, σχιστολιθικό αέριο. Έχουμε μιλήσει για την τεχνολογία μετάβασης. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά και με ανοιχτό μυαλό αυτές τις νέες δυνατότητες. Πρέπει να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις επιπτώσεις για το περιβάλλον, για τους πληθυσμούς, για το ενεργειακό σύστημα και για την οικονομία μας. Είναι σημαντικό επίσης και όσον αφορά τις εκχωρήσεις να υπενθυμίζουμε όσον αφορά τα πυρηνικά και το φυσικό αέριο πρέπει να μην ξεχνάμε τις επιπτώσεις όλων αυτών των ενεργειών. Θα ήθελα λοιπόν να είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα ενδεχόμενα μελετώντας προσεκτικά τις επιπτώσεις και συνέπειες για τους πληθυσμούς και το περιβάλλον και για το συνολικό σύστημα. Ολοκληρώνω εδώ και όταν θα συζητήσουμε ε, για τις τροπολογίες θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να καταλάβουμε ακριβώς ποιες είναι οι επιλογές που θα πρέπει να κάνουμε μέχρι το 2050. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Βαν Το λόγο έχει η κυρία ε, Φιώνα Όλ. Ευχαριστώ. <clears throat> Επικροτώ τον ε, χάρτη πορεία τη Κομισιόν καθώ και τι παρατηρήσει τη εισηγήτρια και ιδιαίτερα την ε, παρατήρηση ότι θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ του ε, τα κράτη-μέλη διότι νομίζω ότι έχουμε κοινά προβλήματα και κοινέ λύσει. Νομίζω ότι ο Χάρτη πορεία είναι θετικό έγγραφο διότι δείχνει ότι η απανθρακοποίηση του ευρωπαϊκού συστήματο ενέργεια δεν είναι μόνο κάτι εφικτό αλλά ότι δεν θα μα τυχήσει και τίποτα παραπάνω από τη συνήθω, διότι μπορούμε να ε, μειώσουμε τις, ε, ενέργειες, τις εισαγωγές ε, καυσίμων μας, το κόστος των οποίων αυξάνεται και έτσι μπορούμε να μειώσουμε το κόστος. Σημαντικό στοιχείο του χάρτη πορείας είναι ότι βρισκόμαστε σε κάποια φάση όπου θα πρέπει να επενδύσουμε σε νέες υποδομές, ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τι σωστέ υποδομέ που θα βοηθήσουν τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Όπω είπε η συγγήτρια, υπάρχουν ε, κάποιε επιλογέ ε, τι οποίε δεν μπορούμε να αποφύγουμε στην έκθεση αυτή. Η απόδοση τη ενέργεια ε, είναι μία από τι επιλογέ αυτέ. τα σχετικά σενάρια δείχνουν ότι μπορούμε να μειώσουμε την ζήτησή μα κατά 41% μέχρι το 2050 σε σχέση με το 2005. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, καθότι εξετάζουμε αυτή τη στιγμή την ε, οδηγία για την ε, ενεργειακή απόδοση. Ε, ο αρχικός μας στόχος είναι μείωση κατά 20% της κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020. Όλα τα σενάρια δείχνουν ε, σημαντική αύξηση στις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γι' αυτό και αυτή είναι μια λύση που δεν μπορούμε να αποφύγουμε ε, στη συνέχεια, που δεν θα πρέπει να μετανιώσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε από αυτό δεδομένου ότι όπως και να το δούμε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, θα πρέπει να παίξουν ε, ε, ρόλο κλειδί. Θα πρέπει να φροντίσουμε ο σχετικός τομέας να έχει τις απαραίτητες επενδύσεις για να προχωρήσει το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τώρα την εκπλήρωση των στόχων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030 η απόδοση της ενέργειας και οι, ε, ανανεώσιμες πηγές, ενέργειας και η απόδοση της ενέργειας αποτελούν δύο στοιχεία τα οποία αν συνδυαστούν μπορούν να μας, δείξουν, να μας φέρουν πολύ καλά αποτέλεσμα ε, και η, ενέργεια που παράγουμε εμείς με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ πιο ε, σίγουρη από αυτήν που θα πρέπει να ε, εισάγουμε. συμφωνώ ότι το αέριο έχει να παίξει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ευελιξία βράχη πρόθεσμα, διότι ότι μπορεί κανείς να, ανάψει κλείσει διακόπτη, να ανοίξει το το διακόπτη, ε, κάτι που διαφέρει από τις ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά το φυσικό αέριο, διότι από τεχνικής πλευράς έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ευέλικτα το φυσικό αέριο και να έχουμε ταυτόχρονα ε, ε, ε δέσμευση και αποθήκευση ε, του άνθρακα. Ε, εάν ε, κάνει κανείς αποθήκευση, δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, καθυστερεί το, το, το, άναμα και το σβήσιμο κάποιες ώρες. Δεν είναι τόσο εύκολο ε, το να ανοίξει ή να κλείσει κανείς το διακόπτη όσο είναι με το ε, φυσικό αέριο. Θα πρέπει να το προσέξουμε λοιπόν αυτό. Εάν θέλουμε φυσικό αέριο θα πρέπει να φροντίσουμε να παραμείνει ευέλικτο και να ε, φροντίσουμε να δημιουργήσουμε υποδομές οι οποίες δεν θα είναι χρήσιμες στο μέλλον. Και συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια ότι μαζί με την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το στοιχείο κλειδί μέχρι το είναι η καλύτερη διασύνθεση. Ε, το να έχουμε τις απαραίτητες υποδομές είναι απολύτως απαραίτητο, αλλά το να έχουμε και το ε, σωστό δίκτυο ε, διανομής είναι πολύ σημαντικό. Σε επίπεδο δικτύου μετάδοσης είναι σημαντικό αυτό. Θα πρέπει να φροντίσουμε η ενεργειακή αγορά να λειτουργεί καλά, αλλά ο πιο φτηνός τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι να πουλάμε και να αγοράζουμε ε, ενέργεια διασυνοριακά. Και η ε, και, υπάρχουν, ε, και υπάρχει και η διάσταση της ε, αποθήκευσης ε, της ενέργειας. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά όπως είναι και τα super grids, τα υπερδίκτυα στην στη Βόρεια Θάλασσα. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να ε, ε, έχουμε ε, ολοκληρωμένα δίκτυα με αιωλική ενέργεια στο βορρά και με φωτοβολταϊκά κύτταρα στον νότο. Έχοντας κατά νου αυτά που είπε η συγγήτρια, νομίζω ότι μας περιμένουν πολύ επικοδομητικές συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στη συνάδελφο Τζόρνταν που είναι σας παρακαλώ να τηρείτε από εδώ και στο εξής τα δύο λεπτά, διότι έχουμε πάρα πολλούς εγγεγραμμένους που θέλουν να μιλήσουν. Έχουν όλοι το δικαίωμα να εκφραστούν, θα χρειαστεί να μοιράσουμε το χρόνο μεταξύ όλων. Παρακαλώ, συνάδελφε. Ωραία, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Και δεν είμαι εισηγήτρια στην ΕΜΒ γιατί είμαι στην Ήτρε τώρα. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας δηλώσω ότι, ότι έχω πρόβλημα. Δεν έχω σλοβενική διερμηνία. Επίσης, ε, συμφωνώ με όσα είπε η συγγήτρια. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη θέση της για την ισορροπημένη προσέγγιση. Σας υποστηρίζω ιδιαίτερα αυτή την ε, ισορροπημένη προσέγγιση που θα πρέπει να αποτυπώνεται επίση και στα όσα λέμε για τις ε, δυνατότητες ε, για τους μελλοντικούς στόχους για το 2030 και όταν μιλάμε για τη στρατηγική για το έτος 2050. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τις τρεις γωνίες του τριγώνου βιωσιμότητας. Εδώ όμως έχουμε κάποιες δυσκολίες. Δεν έχουμε επαρκή δεδομένα στον οδικό χάρτη για το 2050 διότι η Κομισιόν δεν έλαβε υπόψη, η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη και τις τρεις πτυχές της ε, βιωσιμότητας σε ίσο επίπεδο. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα εδώ και θα ήθελα κάποια σχόλια από την Κομισιόν για αυτή την ισορροπία. Το επόμενο θέμα είναι το, η διεθνή πτυχή που είναι κατά την άποψή μου τόσο σημαντική όσο και η εσωτερική ευρωπαϊκή πτυχή διότι αυτός ο δικός χάρτης για την ενέργεια δεν αφορά μόνο την παραγωγή ενέργειας αφορά και τις ενεργειακές τεχνολογίες μας. Και ανησυχώ ότι όλα αυτά τα σενάρια του ενεργειακού οδικού χάρτη θεωρούν δεδομένο ότι υπάρχει παγκόσμια δράση για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα και με τα όσα συμβαίνουν τώρα και στη Βόνη και υπό την Προεδρία της κυρίας Χέντεγκάρντ, χρειαζόμαστε κάποια σενάρια, τουλάχιστον, με, που θα θεωρούν κάτι άλλο δεδομένο. Το επόμενο είναι οι ευθύνε. Πιστεύω ότι ένα έγγραφο σαν αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης και κάποια διάκριση μεταξύ ευθυνών ε, σε ε, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το επόμενο, τα επιπλέον μου σχόλια για τα διάφορα σενάρια είπα ότι όλα τα σενάρια θεωρούν το ίδιο πράγμα δεδομένο, ότι υπάρχει διεθνής δράση για την κλιματική αλλαγή, αλλά δεν παρέχουν ισορροπημένη προσέγγιση για τα αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασία, την εφοδιαστική ασφάλεια και την αλληλεξάρτηση. Το επόμενο σχόλιο για τα σενάρια είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο που λαμβάνει υπόψη τις καθυστερήσεις του CCS και την... το σενάριο low nuclear, χαμηλή πυρηνική ενέργεια προωθείται πολύ σε πολιτικό επίπεδο και είναι πολύ ρεαλιστικό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, ένα σενάριο με το συνδυασμό αυτών των δύο. Επίσης δεν καταλαβαίνω πώς αυτά τα σενάρια λαμβάνουν υπόψη τη συμβατική και τη μη συμβατική χρήση του φυσικού αερίου. Θα ήθελα περισσότερη ολοκλήρωση μεταξύ οδικού χάρτη μεταφορών και ενέργειας. Θα ήθελα να λέγονται περισσότερα για τις εφηδρικές πηγές ενέργειας, διότι τα έξυπνα ενεργειακά σύστημα δεν αφορούν μόνο έξυπνες ρυθμίσεις, αλλά και έξυπνη κατανάλωση και παραγωγή. Επίσης, ε, θα ήθελα να υπάρξουν κάποιες συστάσεις όσον αφορά τη δημόσια αποδοχή που αναφέρεται μόνο ως προϋπόθεση, χωρίς καμία άλλη σύσταση στην έκθεση της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ο χρόνος είναι αυτός που είναι και δεν περνάει πολύ γρήγορα. Κύριε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η απάντησή μου θα είναι πολύ σύντομη. Ήθελα να πω περισσότερα πράγματα, αλλά δεδομένων των χρονικών περιορισμών θα ε, παραμείνω στην ανάλυση των σενάριων. Πρέπει να πω ότι τα το κυριότερο σενάριο, αυτό που αφορά την ενεργειακή απόδοση, μου φαίνεται εξάλλου όπως ε, αναφέρεται και στην έκθεση του κ. Τόμς, είναι εσφαλμένη η έκθεση θα έλεγα διότι συγχαίει το μέσο με το στόχο. Πιστεύω επίσης ότι η εξοικονόμηση, η απόδοση βρίσκεται σε επίπεδο παραγωγής, συνεπώς στην πλευρά της ενεργειακής βιομηχανίας και όχι όπως θέλει η Κομισιόν και ο κ. Τζόμπς ε, στην πλευρά των καταναλωτών. Τέλος, πιστεύω η Κομισιόν παραβλέπει τον άνθρακα, το κάρβουνο. Δεν μιλάμε για το αέριο που προέρχεται από διαδικασίες υψηλής θερμοκρασίας. Σε αυτό το σενάριο δεν λέμε τίποτα για τη θερμική ενέργεια. Υπάρχει, υπάρχουν σήμερα τεχνολογίες που επιτρέπουν να, μειώσουμε τη θερμοκρασία σε αυτή. Λοιπόν, η φυσική αντιδραστήρα, αυτός ο φυσικός αντιδραστήρας που είναι η γη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα μπορούσαμε να πάμε σε μεγάλα βάθη και να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια που υπάρχει εκεί πέρα στο βάθος. Πρόκειται για μια τεχνολογία για το μέλλον της Ευρώπης μεταξύ άλλων. Υπάρχουν χώρες όπως η Τουρκία Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε που ήσασταν πολύ σύντομος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν κοιτάξουμε τον ε, χάρτη πορείας, ε, βλέπουμε ότι μας ε, δίνει μια ιδέα του πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε θέσεις πάνω σε σημαντικές στατικές πέρα από το έτος 2020 που είναι ο πιο κοντινός μας ορίζοντας. Καταλαβαίνω ότι για πολλούς ε, συναδέρφους αυτές οι μακροπρόθεσμες ε, πρόπτικες οδηγούν ε, σε κάποιο σκεπτικισμό διότι υπάρχουν πολύ άγνωστοι παράγοντες όταν μιλάμε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν μιλάμε όμως για την ενεργειακή πολιτική, οι υποδομές απαιτούν αρκετό χρόνο για να δημιουργηθούν, και χρειάζεται αρκετός χρόνος ε, μέχρι να μπορεί κανείς να επωφεληθεί ε, από τις επενδύσεις που έχει κάνει. Και Βλέπουμε ότι οι υποδομές μας είναι αρκετά παλιές ε, όσον αφορά το, τον αναμενόμενο κύκλο ζωής τους. Ε, θα πρέπει λοιπόν να είμαστε φιλόδοξοι όταν ε, κοιτάμε αυτές τις διάφορες πτυχές. Η Κομισιόν έχει παρουσιάσει μια σειρά ιδεών που αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε, ιδιαίτερα όταν... Και γι' αυτό θα στηρίξουμε την προσπάθεια για ενεργειακή αποτελεσματικότητα, να έχουμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση στην αγορά, κάτι το οποίο μας οδηγεί ε, στο να μην έχουμε πια ενεργειακές νήσους, να δούμε τι θα γίνει με το μη συμβατικό φυσικό αέριο και αυτό είναι πάρα πολύ στο προοπτική, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε το ισχύον πλαίσιο αναφορά, να δούμε τι θα κάνουμε με ένα μείγμα ενεργείου που να περιλαμβάνει την πυρηνική ενέργεια και τελικά να απαλλαγούμε από τις βλαπτικές ε, εκπομπές αλλά επίσης να δούμε και το ότι αυτό που χρειάζεται είναι το πώς θα περιορίσουμε, τουλάχιστον να κρατήσουμε μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, το, το, το, κόστος και την ε, τιμή. Επίσης, να δούμε τι θα γίνει με τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Κάτι το οποίο αφορά το πόσο έχουμε προχωρήσει όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μη συνεχείς ε, μορφές ενέργειας, να δούμε τι θα γίνει ε, ε, με τις μορφές ενέργειας που δεν μας οδηγούν σε εκπομπές διοξιδίου. Θέλουμε επομένω μια υγιή αγορά και όχι μια αγορά που έχει τα δεκανίκια των επιδοτήσεων, κάτι το οποίο δεν έχει μέλλον. Επίσης θα πρέπει να δούμε αυτό το οποίο είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε το πώς οι τιμές θα αντικατοπτρίζουν το κόστος με περισσότερη πιστότητα και ακρίβεια. Και επίσης να δούμε πώς θα έχουμε τις ε, σχετικές επενδύσεις. Και επίσης να δούμε κάτι το οποίο το ε, λέμε εδώ και καιρό, το ότι, το πώς ε, θα αποφύγουμε της, την τεχνητή διαμόρφωση που, των τιμών που φέρνει μία στρέβλωση στην αγορά, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και επίσης να δούμε το ότι έτσι αποθαρρύνεται και η αποταμίευση και η ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Να σταματήσουμε τη μικροπολιτική και τις, τις προεκλογικές κραυγές και θα πρέπει επομένω να προσγειωθούμε, να είμαστε ρεαλιστές γιατί να δούμε το ότι η κρίση προβληματίζει και είναι σωστό αυτό. Θα πρέπει να μην δίνεται έτσι όθηση προς τα πάνω για τις τιμές. Χρειάζεται επομένω ένας χάρτης πορείας. Και θα πρέπει αφενός να έχουμε ένα μακρόπνομο προγραμματισμό, αφετέρου όμως να μην ξεχνούμε τη σημερινή συγκυρία. Άρα, έτσι, κρυστάλλινη θέση να υιοθετήσουμε για το μέλλον της ενέργειας και να δούμε το πώς θα προλιάνουμε το έδαφος ούτω ώστε οι σχετικές νομοθετικέ προτάσεις να πάνε καλά για τα μέσα επόμενα χρόνια. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βομπίσκα. Σας ευχαριστώ. Προσπαθούμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον της ενέργειας, να είμαστε έτοιμοι, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτού που επενδύουν στον κλάδο. Όλα συνεχώ αλλάζουν. Θα πρέπει εμεί και εμεί να έχουμε κάποιου στόχους μακρόπνοους και επίσης να δούμε το πώς θα έχουμε κάποια πολιτική που θα περιορίζει τις εκπομπές διοξιδίου. Τέτοιο χαρτί πορείας θα πρέπει να φτιάξουμε. Φτάνουμε στο 90% της ενέργειας που παράγεται σε κάποια χώρα που θα πρέπει να αλλάξει προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Κάτι άλλο τώρα. Το πώς θα μπορέσουμε τελικά να ελοπίσουμε τους στόχους που έχουμε τάξει. Γιατί δεν αρκεί να τάσει κανείς στόχους. Θα πρέπει και να τους υλοποιεί. Θα πρέπει επομένως να υπάρχει εποπτεία και παρακολούθηση του αν τηρούνται οι κανόνες που έχουμε θεσπίσει. Επίσης, η κάθε χώρα να έχει το δικό τους χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για γενικούς πανευρωπαϊκούς χάρτες πορείας. Όμως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσαρμόζουμε αυτά τα οποία απαιτούμε εις τις ιδιοτροπίες, ιδιορυθμίες κάθε χώρας. Να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες σε συγκεκριμένα σημεία. Κάτι τελευταίο τώρα. Από όσα άκουσα από τους συναδέλφους, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής. Να λάβουμε υπόψη τις μελέτες που έχουν γίνει αλλά και τις εκθέσεις που έχουν γίνει για το φυσικό αέριο. Στην Ήτρε ε, υπάρχει κάποια συνάδελφος που συντάσσει τώρα κάποια έκθεση από την οποία θα μπορούσαμε να δανειστούμε πολύτιμες πληροφορίες. Είναι και θέμα ενεργειακής ασφάλειας. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν. Έχουμε επίσης και το θέμα της ε, διεθνού αρχής, της διεθνούς υπηρεσίας για την ενέργεια. Να δούμε τι θα γίνει με... Ναι. Τι mm, e, θα γίνει με την e, δέσμευση, τι θα γίνει με την e, αποθήκευση του διοξιδίου. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το κύριο Δεν θα μακρηγορήσω γιατί τα είπαμε και θα περιοριστώ στα εξή λίγα. Ε, πάρα πολύ θετικά τα όσα μας είπε η συγκήτρια για την ενεργειακή ασφάλεια. Είναι κάτι το οποίο δεν με απασχολεί γιατί δεν είναι το θέμα του πώς θα απαλλαγούμε από το διοξίδιο αλλά πώς θα πετύχουμε ενεργειακή ασφάλεια γιατί είναι και θέμα έτσι εθνικής ασφάλειας. Αυτό χρειάζεται ο κόσμος. Αυτό θα το πετύχουμε μειώνοντας τις ενεργειακές ανάγκες αλλά και αυξάνοντας την ενεργειακή ασφάλεια. Η σταχτοπούτα το, της, της ασκούμενης πολιτικής μας είναι το θέμα αυτό. Βέβαια και είναι πολύ εύστοχη η προσέγγιση της ε, Επιτροπής, μπράβο της όσον αφορά τους χάρτες πορείας. Νομίζω ότι καμιά φορά ε, είναι πιο αποτελεσματικοί οι τεχνοκράτες από τους πολιτικούς. Και έτσι και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουν τα κρατημέλη που φυσικά δεν να πάρουν τις ε, αποφάσεις τους. Εμείς, ξέρετε, στη σκοτία κάνουμε ό,τι ό,τι μπορούμε όσον αφορά <clears throat> έχουμε και αυτή την λοταρία όπως τη λέμε την ενεργειακή και θα πρέπει να δούμε τι ζητούν οι αγορές το είπαμε και σε σχέση και με το πακέτο των έργων υποδομής ακόμα δεν πετύχαμε μια πραγματικά ενιαία αγορά και αυτό είναι κακό και για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, αλλά θα πρέπει να δίνουμε τις προσπάθειές μας και όσον αφορά τα έργα υποδομής και όσον αφορά επίσης τις νομοθετικές ρυθμίσεις που να σταματήσουν να είναι τροχοπέδια. Θεωρούμε ότι η ενέργεια θα πρέπει να παραμείνει εθνική αρμοδιότητα. Όμως, τα πιο πολλά θα πετύχουμε συνεργασία παρά εάν έχουμε ο καθένας ξεχωριστές προσπάθειες. Έμεινα στο χρονικά πλαίσιο που μου ζητήσατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα δευτερόλεπτα αφήσετε, συνάδελφε βέβαια. Θα προσπαθήσω να είμαι το ίδιο σύντομο, θα περιοριστώ σε ένα μόνο σημείο. Αυτή η εξαιρετική έκθεση αναφέρει τέσσερις ε, φορείς, τέσσερις άξονες για τη μείωση του άνθρακα και ο τρίτος από αυτούς τους παράγοντες είναι η πυρηνική ενέργεια. Πιστεύω ότι αυτό είναι εξαιρετικό, διότι δεν υπάρχει τρόπος να επιτύχουμε το στόχο της μείωσης των εκπομπών άνθρακα εάν εγκαταλείψουμε την πυρηνική ενέργεια. Μπορεί να μην μας αρέσει, Ξέρουμε ότι αυτή η ενέργεια έχει υψηλό κίνδυνο, η καταστροφή της Φουκουσίμα μας το υπενθυμίζει αλλά δεν υπάρχει ενέργεια που μπορεί να την αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή και στο προβλέψιμο μέλλον. Δεν μπορούμε λοιπόν να δρούμε χωρίς αυτήν. Αυτή η έκθεση το λαμβάνει υπόψη και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ξέπαινο. Δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτήν εκτός ε, εάν ε, ανατρέξουμε ε, μαζικά στον άνθρακα, στο πετρέλαιο, στο σχιστολιθικό αέριο που έχουν μεγάλες εκπομπές ε, και πολλούς ρήπους και που έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους μας για τη μείωση του άνθρακα. Εφόσον λοιπόν λάβουμε υπόψη αυτό το τρίτο παράγοντα, το κεντρικό ερώτημα είναι, το κεντρικό ζήτημα είναι η μείωση, η ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτού του τύπου ενέργειας. Αυτό συνεπάγεται επενδύσεις δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν σήμερα στα κέντρα παραγωγής ε, πυρηνικής ενέργειας. Ε, πρέπει να επενδύσουμε στη νέα γενιά, στην τέταρτη, στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, στο παροπλισμό που μπορεί να αποτελέσει μια ευρωπαϊκή βιομηχανία, διότι τα πυρηνικά επεκτείνονται στο στον κόσμο, η Ινδία, η Κίνα ε, χρησιμοποιούν και αυτή και αυτές οι χώρες αυτή την ενέργεια και δεν μπορούν να την εγκαταλείψουν. Το ζήτημα λοιπόν της ασφάλειας, των εγκαταστάσεων αυτών, της επεξεργασίας των αποβλήτων, του παροπλισμού θα ε, μπορούσε να αποτελέσει μια βιομηχανία στην οποία θα μπορούσαμε να αριστεύσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια δυναμική θέση για την αντιμετώπιση αυτής της νέας μορφής, ε, μεταβατικής μορφής ενέργειας, μεταβατικής αλλά απαραίτητης. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε την έκθεση αυτή κυρίως για το μέλλον, για τα επόμενα 30 χρόνια όσον αφορά αυτή την ενέργεια. Ευχαριστούμε τον συναδελφό Βέμπερ. Το λόγο έχει η κυρία Ζουδίτ Μέρκες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Πρέπει να πω ότι όσον αφορά του οδικούς χάρτες συνήθως ξεκινάμε από μια πραγματική κατάσταση ε, ωστόσο τα πράγματα δεν θα είναι τα ίδια το 2050. Πιθανώς τότε θα χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια. Εμείς ξεκινάμε με τα σημερινά δεδομένα. Σκεφτόμαστε ότι πρέπει να περάσουμε από τον άνθρακα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια άριστη ιδέα, ωστόσο γνωρίζουμε ότι το μέλλον είναι μια υπόθεση που κάνουμε βάσει των σημερινών ε, συνθήκων. Θα χρειαστεί ωστόσο να σκεφτούμε και ε, μεγάλη σειρά διαφόρων λύσεων. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε θεωρώντας δεδομένη τη σημερινή παραγωγή ενέργειας με τις εγκαταστάσεις που έχουμε σήμερα το 2050. Ίσως θα, βρεθούμε, θα βρισκόμαστε σε διαφορετική κατάσταση πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε ίσως ενδεχομένως κάθε πολίτης να μπορεί να παράγει τη δική του ενέργεια μέσω παράδειγμα ηλιακών συλλεκτών ώστε να είμαστε ακόμη πιο αποδοτικοί αξιοποιώντας ε, και ανακυκλώνοντας το ζωστό νερό και ούτω καθεξής. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δείξουμε θάρρος, θα πρέπει να σκεφτούμε τη μικροενέργεια, το τι μπορούν να παράγουν οι επιμέρους πολίτες. Εάν δράσει έτσι ο πολίτης ε, και επιτευχθεί μέσω των επιχειρήσεων να αξιοποιηθούν ε, τα υπόλοιπα ενέργειας θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτό σήμερα δεν γίνεται επαρκώς. Πρέπει να πω ότι η έκθεση αυτή προς το 2050 είναι πολύ καλή αλλά θα ήθελα να απευθυνθώ στην εισηγήτρια και να της πω ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να είναι λίγο πιο επικοδομητική όσον αφορά το 2050. Ευχαριστούμε πολύ και που τηρήσετε το χρονικό όριο. Το ρόλο έχει ο Βιτσέντσο. Κύριε Βιτσέντσο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται ότι οι σοσιαλιστές είναι πολύ δραστήριοι σήμερα. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα που... Είπα το να μιλάμε πολύ δεν σημαίνει ότι είμαστε δραστήριοι για να σας πω ένα λόγο, να σας πω κάτι. Ε, όλοι έχουν διατηρήσει τη ε, χρονικά όρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και την Κομισιόν για την προετοιμασία αυτού του σχεδίου. Μας δείχνει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι επίτευξης του ίδιου αποτελέσματος και πιθανώς το 2050 στην Ευρώπη, σε κάθε περιοχή θα υπάρχει ίσως μια λύση πολύ διαφορετική από αυτή που προσφέρεται σήμερα ο δικός χάρτης λοιπόν θα είναι συνδυασμό των διαφορών σεναρίων σε άλλες χώρες θα υπάρχουν πυρηνικά σε άλλες θα υπάρχουν, έχουν, έχουμε άνθρακα και σε άλλες έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτό που με φαίνεται πιο ενδιαφέρον ότι θα πρέπει να Πάμε πέρα από αυτό το διάλογο για τις πιθανούς πόρους για το 2050. Διάβάστε προσεκτικά το έγγραφο, θα δείτε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ότι από το 10% του ΑΕΠ σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ενέργεια θα αυξηθεί στο 14% το οποίο σημαίνει αύξηση τουλάχιστον 40% του ενεργειακού τομέα στο ΑΕΠ. Δηλαδή θα είναι οι κεφαλιακές δαπάνες πολύ υψηλότερες, υψηλότερες σε σχέση με τις αυξομοιούμενες τιμές που έχουμε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα διότι όλο αυτό αφορά τις πιθανές επενδύσεις. Αυτό το επενδυτικό σχέδιο μαζί με την υπόλοιπη νομοθεσία που θα συζητήσουμε σήμερα και που θα συζητήσουμε στο μέλλον πιστεύω ότι κάποια ζητήματα πρέπει να συζητηθούν περισσότερο σε βάθος. Ε, οι τιμές του διοξιδίου του άνθρακα για το μέλλον θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πιστεύω και ίσως να αυξηθούν ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί αυτό εδώ, διότι θα αποτελέσει μία από τις κινητήριες δυνάμεις για τους πιθανούς επενδυτές ώστε να συμμετέχουν στις περιφέρειες. Αυτή είναι λοιπόν μια συζήτηση που θα πρέπει να κάνουμε ξεχωριστά στην επόμενη συζήτησή μας και σίγουρα η δημόσια αποδοχή που συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τη δημόσια αποδοχή των διαφορών αλλά και των τιμών των ενεργειών και τιμών με τις οποίες πολλούνται στους καταναλωτές και το μισό εκατομμύριο Ευρωπαίοι κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενέργεια αυτή και αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση για μας και πρέπει και αυτό να περιγράφεται καλύτερα στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Mm, ε, ε, ε, Έλμερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον κύριο Βέμπερα Ναι, θα πρέπει να είμαστε υπέρ τη πυρηνική ενέργεια που θα μα βοηθήσει στο μέλλον. Και κάθε φορά που ε, μιλάμε για την πυρηνική ενέργεια, αρχίζουμε και απολογούμε θα ταυτόχρονα και για την ασφάλεια. Για κοιτάξτε τι γίνεται με του δείκτε θνησιμότητο. Ε, Α πούμε στην, στον τομέα και στο, στον τομέα που χρησιμοποιεί τον άνθρακα. Όχι. Είναι, είναι, είναι κατά, πολύ, κατά, κατά πολλέ τάξει μεγέθους ασφαλέστερη η πυρηνική ενέργεια. Τώρα, ε, θα ήθελα να πω στην κυρία Χόλ το εξή. Διαφωνώ. Εκεί που είπατε ότι η ενέργεια από τι ανανεώσιμε είναι πιο ασφαλέστερη ε, παρά η εισαγωμένη ενέργεια. Δυστυχώ τα ανανεώσιμα είναι απρόβλεπτα. Δεν είναι συνεχού ε, μορφή. Ε, δεν είναι να θεωρηθούν ασφαλεί πηγέ ενέργεια όσο εφάνταστο και να είναι κανεί. Βεβαίω είναι δυνατόν κανένα να έχει ενέργεια μέσω της χρήσης του νερού, θεωρητικά, όμως δεν έχουμε τη δυνατότητα ε, να αποθηκεύσουμε από όλες τις ενενώσιμες πηγές ενέργειας της Ευρώπης. Ε, δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε και μας είπε επίσης ότι οι αγοραπολισίες μεταξύ των χωρών θα βοηθούσαν, ε, όμως είδατε τι έγινε. δεν, δεν, δεν, δεν λείπει ο ήλιος μόνο τη Σκανδιναβία, πολλές φορές λείπει και από την Ιταλία. τι να κάνουμε στην Ευρώπη, πολλές φορές υπάρχει τέτοιο συντονισμός και ούτε και αυτό που λένε οι πράσινοι ότι παντού υπάρχει αέρας. Όχι, πάρα πολλές φορές υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη που υπάρχει άπνοια. Οπότε, ε, κατά αυτόν τον τρόπο, κάποιος χρειάζεται τον backup, δεν μπορεί να, να στηρίζεται σε ήλιο και άνεμο. Το, θέμα είναι βέβαια ότι πολλές φορές έχουμε ε, τις ανανεώσιμες, αλλά δεν έχουμε το φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να ε, είναι η εναλλακτική πηγή σε, περίπτωση ανάγκης, στον backup. Ε, γι' αυτό σας λέω, ε, προσοχή, υπάρχουν κάποια προβλήματα όπως έχουν εμφανιστεί στη Γερμανία, γιατί με πάρα πολλές πράσινες πολιτικές καταστρέφουν την ενεργεία μας πολιτική ουσιαστικά. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα η εκπρόσωπος της Κομισιόν, κ. Βορσόφ, από την οποία θα ζητήσω να μην μιλήσει περισσότερο από δύο λεπτά αν έχει την καλοσύνη. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια την κυρία Τσαβέλα. Ευχαριστώ και όλους ε, τους βουλευτές που πήραν το λόγο. Κάποιες παρατηρήσεις για τον ενεργειακό χαρτί πορείας για το 2050. Βασικά συμφωνούμε με όλα όσα υπόθηκαν και που προτείνατε να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Πράγματι, ο ενεργειακός ε, χάρτης πορείας ε, για το 2050 στόχο έχει να καθοδηγήσει τις ε, κυβερνήσεις. Δεν προβλέπουμε το μέλλον, έχουμε κάνει κάποιες υποθέσεις, γνωρίζουμε πολύ καλά την αβεβαιότητα που υπάρχει και στόχος είναι περισσότερο να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ε, γνωρίζετε ότι τα διάφορα σενάρια μας βοηθάνε να καταλάβουμε τι θα γίνει εάν ακολουθήσουμε τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε τους τρεις στόχους ε, της ενεργειακής πολιτικής αηφορία, ασφάλεια τροφοδοσίας και ενεργειακή απόδοση. Ε, έχουμε κοιτάξει τα διάφορα σενάρια, έχουμε εξετάσει ε, τα διάφορα θέματα του κόστους ε, και έχουμε συγκρίνει το κόστος. Και από τα διάφορα σενάρια αυτά και από τη δουλειά ενδιαφερομένων κύκλων και κρατών μελών ε, καταλήγουμε στο ότι όλοι συμφωνούμε ε, σε αυτές τις τρεις ε, απαραίτητες λύσεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υποδομές και όπως σας είπα, τα σενάρια αυτά δεν αποτελούν προβλέψεις, μας βοηθάνε να συγκρίνουμε τις διάφορες επιλογές, μας δίνουν πράγματα να σκεφτούμε και υπάρχει και η μελέτη επιπτώσεων που συνοδεύει τον χάρτη πορείας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας ρώτησε πέρυσι τον Φεβρουάριο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συμφωνία, το deal, ε, και μας ρώτησαν επίσης τι θα γίνει εάν η ε, Ευρωπαϊκή Κοινότητα ε, ενεργήσει μόνη της και αυτό καλύπτεται στον χάρτη πορείας. Επίσης έχουμε συνεργαστεί στενά σε επίπεδο σε επίπεδο επιτροπής ε, και με άλλους ε, τομείς της Επιτροπής. Ε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουμε συμπεριλάβει στο σενάριο. Το ένα είναι το αέριο από σχιστόλιθο. Είναι αρκετά βέβαιο το θέμα αυτό. Εξετάζουμε το θέμα στο έγγραφο πολιτικής και όπως σας και καθότι δεν έχω πολύ χρόνο, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειε των διαφόρων ε, ενεργειακών πόρων. Ε, όπω είπαμε, όλοι οι πόροι είναι σημαντικοί. Σημαντικό είναι τώρα να καθορίσουμε το πλαίσιο πολιτική για το 2030 και ο χάρτης ε, πορεία στόχο έχει να βοηθήσει στον καθορισμό των στόχων για το 2030. Ευχαριστώ. Είναι λίγο συνήθιστο, έχουμε κλείσει τον κατάλογο και ο συνάδελφος Μεζάρος μας ζητάει να μιλήσει. Παρακαλώ πραγματικά μισό με πολύ, το πολύ ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα τις παρατηρήσεις. Δεν ζήτησα το λόγο... Ζήτησα το λόγο γιατί θέλω να δω κατά πόσο το πρόγραμμα ITER ε, αποτελεί κομμάτι του εγγράφου, διότι πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο και ήθελα να προτείνω. Ζητώ συγγνώμη, η γραμμάτια μου είπε ότι κουνήσατε το καρτελάκι και έτσι ζητάτε το λόγο. το... Ζήτησα το λόγο, όντως, κυρία Πρόεδρε. Ξεκίνησα να μιλάω, πήρα το λόγο, ήθελα να πω κάτι, κυρία Πρόεδρε. Μπορώ να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, κυρία Πρόεδρε. Είπατε δεν ζήτησα το λόγο και έτσι κατάλαβα ότι δεν ζητήσατε το λόγο. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε πολύ σύντομα γιατί ούτως ή άλλως είχε ολοκλη... Ε, κλείσει ο κατάλογος. Την επόμενη φορά θα μιλήσω στα αγγλικά, ίσως θα είναι πιο απλό. Λοιπόν, εν συντομία, παίρνω το λόγο σε αυτό το σημείο διότι διάβασα λίγο το έγγραφο για να δω κατά πόσο το πρόγραμμα ITER εντάσσεται σε αυτό αλλά πόσο είδα δεν αναφέρεται το πρόγραμμα ITER. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν να τη ζητήσω να λάβει υπόψη αυτό το πρόγραμμα ITER σε αυτό το έγγραφο διότι το 2026 το πρώτο κέντρο παραγωγής θα τεθεί σε λειτουργία και τη δεκαετία του 30 το πρόγραμμα ITER θα παράγει ενέργεια. Θα πρέπει λοιπόν το πρόγραμμα ITER να ε, αποτελεί κομμάτι αυτού εδώ. Ωραία, για να ολοκληρώσουμε ζητάω την κυρία Τζαβέλα να μιλήσετε εν συντομία. Σας υπενθυμίζω ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες πρώτα απ' όλα όταν θα συζητηθεί η έκθεσή σας που, την οποία θα μας παρουσιάσετε 11-12 Ιουλίου. Με εκείνη την ευκαιρία θα ξαναμελετήσουμε όλα τα θέματα. Στη συνέχεια οι συντονιστές σκέφτονται μία δημόσια ακρόαση που θα διοργανωθεί και μετά από αυτή την ακρόαση θα έχουμε την προθεσμία για τις τροπολογίες, πιστεύω το Σεπτέμβριο και μετά. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ τώρα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, το λέω για να σας ζητήσω συγγνώμη για όσους θέλαν να προσθέσουν και άλλα. Επειδή βιαζόμαστε, σας ζητώ, κλείνω τη συζήτηση και ζητώ σε εσάς συνάδελφε να ολοκληρώσετε. Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων, θα ακολουθήσουν και άλλες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την συνεισφορά τους σε αυτή τη συζήτηση. Σημείο πρώτο, ε, από τα σχόλια κρίνω ότι η, το, η αναφορά βρίσκεται σε καλό δρόμο. δηλαδή περίπου ό,τι ελέγχθη πράγματι συμπεριλαμβάνεται. Δεύτερο σημείο, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι η αναφορά θα κινηθεί μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Βιομηχανία, Ενέργεια και Έρευνα και Τεχνολογία. Και έτσι ελπίζω ότι θα είμαστε πιο επικοδομητικοί. Και τρίτον, γενικά θα έλεγα ότι μέσα στο πλαίσιο του 2030, της πολιτικής 2030, αυτό το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι έναν γενικό χάρτη πορείας όσον αφορά την ενέργεια για τους πολίτες, τις κυβερνήσεις και την αγορά στην Ευρώπη και διεθνώς. Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο στο χρονοδιάγραμμα και να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι ε, το απόγευμα στη συνάντηση των συντονιστών θα ζητήσω μία κρόαση για αυτό το θέμα γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έπρεπε να κάνουμε μία ακρόαση για να ακούσουμε και τις ε, απόψεις των μετόχων επί του θέματος αυτού. Ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ τη συνάδελφο κυρία Τζαβέλα που ήταν σύντομη. Όπως είπα πριν σας δώσω το λόγο, αυτή είναι μια απόφαση που θα λάβουν οι συντονιστές της σημερινής συνεδρία και είμαι σίγουρη ότι δεν έχουν καμία αντίρρηση γι' αυτό. Μετά τη συζήτηση λοιπόν της έκθεσής σας, της πρότασής σας, 11 και 12 Ιουλίου, Πιθανότατα το Σεπτέμβριο θα λάβει χώρα αυτή η δημοσία κρόαση δεδομένη τη σπουδαιότητα του ζητήματο. Ευχαριστώ όλου. Το επόμενο σημείο αφορά την παρουσίαση εκ μέρου τη ε, Επιτροπή. Ελπίζω όσοι φύγετε να φύγετε χωρί να κάνετε πολύ φασαρία. Παρουσίαση λοιπόν της πρότασης εκ μέρους της Επιτροπής μιας πρότασης για μια ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομία σχετικά με τις πρώτες ύλες. Έχουμε μόλις 30 λεπτά για ολόκληρη τη συζήτηση. Ζητώ από τον κύριο Κοτζιγκού που μας παρουσιάζει αυτή την έκθεση να περιοριστεί σε 10 λεπτά και όχι περισσότερο. Ευχαριστώ. Merci Madame Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι... Παρακαλώ, οι συζητήσεις μπορούν να συνεχιστούν εκτός της αιθούσης. Ευχαριστώ. Εάν έχετε να συζητήσετε, μπορείτε να βγείτε. Μπορείτε να πείτε στην κυρία και στον κύριο, παρακαλώ, να... Thank you for the opportunity to... Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που δώσατε να παρουσιάσουμε αυτή την πρόταση που αφορά τις πρώτες ύλες. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε και πάλι το πόσο σημαντικές είναι οι πρώτες ύλες. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 και το 2011 έχει δημοσιεύσει τι σχετικές ανακοινώσεις. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, μπορείτε να περάσετε έξω, λέει πρόεδρος σε αγγλικά και γαλλικά. Επαναλαμβάνει λοιπόν ο μιλητή, είναι σημαντικέ οι πρώτε ύλε, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Έχουμε αυτέ τι δύο ανακοινώσει το 2008 και 2011. Τότε συγκροτήθηκε και εφαρμόστηκε η σχετική μας στρατηγική. Το 2010 ετοιμάσαμε την ανακοίνωση του 2011 και επίσης ε, ετοιμάσαμε την πρωτοβουλία για το 2020. Τότε επομένω διαμορφώθηκε αυτή μα η σύλληψη. Τι είπατε, τι είπατε, κάποιο ρωτάει από κάτω χωρί μικρόφωνο. Και οι δυνατότητες καινοτομίας υπάρχουν και είναι σημαντικές για πολλές πρώτες ύλες. Ανέκαθεν πιστεύαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις πρωτεσίλες και σε χαμηλές τιμές. Αυτό βέβαια δεν ισχύει πάντοτε. Ε, λείψαν πάντως οι επενδύσεις. Κάποιοι περιορισμοί σε εξαγωγές από τις χώρες που το παράγουν και χειρονοτομία θα έπρεπε να συμπιέσει τις τιμές και από πλευράς προσφοράς μπορούμε να έχουμε καινοτόμες λύσεις, λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία και όσον αφορά την εξόρυξη και την εκμετάλλευση και την επεξεργασία. Επίσης, από πλευρά ζήτηση χρειάζεται ανακύκλωση αποτελεσματική, το οποίο πάντοτε βοηθά, όπως και ο σχεδιασμός των προϊόντων. Και αυτό βοηθά και έτσι μπορούμε να ανακτήσουμε πρωτογενείς ή δευτερογενείς πρώτες ύλες. και να αναπτύξουμε ό,τι χρειάζεται και επίση με τυποποίηση και επιστοποίηση. Όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν και να ενθαρρυνθούν. Τρεις είναι εμπλεκόμενοι στην καινοτομία, τρεις μεταβλητές Πολλές φορές λείπει η γνώση, λείπουν οι επαφές μεταξύ των παραγωγών πρώτων μελών. Συνεργασία μεταξύ των πρώτων μελών. Ας πούμε γεωλογικές έρευνες γίνονται, αλλά δεν υπάρχει συμβατότητα τόσο να υπάρχει ανταλλαγή των πληροφοριών. Η έρευνα στην Ευρώπη, επομένως, είναι ε, κατευθυνμένη. Το 2004 είπαμε ότι ξεκινάει μια εταιρική σχέση για την ε, καινοτομία και χαιρετήσαμε και το ψήφισμά σας του Σεπτεμβρίου που ήταν υπέρ της πρωτοβουλίας μας. Το Φεβρουάριο, γιατί βάσαμε τη σχετική πρόταση, με στόχο να γίνει πρωτοπόρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετάλλευση, επεξεργασία, ανάκτηση κλπ. Πάρα πολύ βασική στόχη που τάξαμε σε αυτούς του τρεις πυλώνες. Από της πρόσφορας και εντός και εκτός της Ευρώπης. Και επίσης το τι θα γίνει με την ανακύκλωση και τις πρώτες ύλες καινοτομία. Επομένω, εκτό από την έρευνα, είναι κάτι το οποίο μα δίνει μια προσέγγιση και δίνει και λύση στην αγορά. Ο ορίζον του 2020 είναι το, ε, και, το, και το πρόγραμμα πλαίσιο, υπαριθμόν 8. Πρόκειται για αυτές τις προκλήσεις αυτές που έχουν διατυπωθεί σε αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο, τι θα γίνει με την κλιματική αλλαγή, θα γίνει με τις πρώτες ύλες, είναι όλα αυτά τα θέματα τα οποία ε, είναι υλοσυνδεδεμένα. Και οι πρώτες ύλες βέβαια είναι από τα πιο βασικά θέματα. Συμμετοχή της βιομηχανίας και κατακλείδη θα πρέπει να σας πω κάτι πρώτα πρώτα όσον αφορά το χρονισμό, το timing, ότι η επόμενη φάση είναι το ότι ελπίζουμε το Συμβούλιο να εγκρίνει τον Δεκέμβριο με τα συμπεράσματά του την ε, πρότασή μας. Κάτι το οποίο δεν έγινε προηγουμένως και ελπίζουμε ότι με την Κυπριακή Προεδρία θα πετύχουμε αυτό και ότι θα, είναι πρόσδετες θα πιάσουν τόπο οι προτάσει μα. Ε, Όμω δεν χάνουμε χρόνο μεταξύ. Ήδη έχουμε αρχίσει την προπαρασκευή. Ο κ. Μπουτικόφερ είναι εδώ και ξέρει τι κάνουμε με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Κάναμε αυτό ακριβώς που είχατε προτείνει και εσείς, το είχατε ζητήσει. Και όσον βρω τώρα καθ' αυτή την εταιρική σχέση της ε, καινοτομίας έχουμε μια ομάδα υψηλού επίπεδου που διατυπώνει συμβουλές, προτάσεις, κατευθυντήριε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το 2013 του χρόνου και προβλέπουμε συμμετοχή να καταναλώσει επίπεδο υπουργών να συμμετάσχει ο κλάδο, ο βιομηχανικό, οι μη κυβερνικές οργανώσεις και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οπότε, πάρα πολύ σύντομα, θα κάνουμε ένα διαγωνισμό για όλους τους ενδιαφερομένου. και να, αυτό είναι χειροπιαστή απόδειξη ότι προχωρεί η υπόθεση. Όμως χρειαζόμαστε πρώτα-πρώτα να, δώσουμε, να το Συμβούλιο το πράσινο φως. Θα έχουμε τους Σέρπα που θα βοηθούν την ομάδα υψηλού επίπεδου. Πέντε επιχειρησιακές ομάδες. Τεχνοκρατική και μη τεχνοκρατική προσέγγιση για επεξεργασία, ανακύκλωση, για την υποκατάσταση, για ε, τα υλικά αυτοκινητοβιομηχανίας. Ε, η ομάδα 3 και 4 δεν θα έχει τεχνολογικό χαρακτήρα θα αφορά τις υποδομές ε, γνώσης, δηλαδή δεξιότητες, δεδομένα κλπ. Και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας επίσης πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία. Το 2014 όσον αφορά τις πρώτες ύλες. Επομένως και η τέταρτη ε, ομάδα εργασίας θα αφορά την ανακύκλωση, θα έρχονται την ανακύκλωση, τους διαγωνισμούς, του κρατικές προμήθειες, ούτως ώστε η ανακύκλωση να γίνει πιο οικονομική. Αυτό θα γίνει με πιο αποτελεσματική συλλογή των απορριμμάτων. Θα εξεταστεί επίση το πώ θα μπορέσει να βοηθήσει η πιστοποίηση και η τυποποίηση και η τελευταία ομάδα εργασία θα σου με το πώς μπορούμε να συντονίσουμε τι προσπάθειέ μας για να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τι πρώτες Οπότε δουλεύουμε εν αναμονή των αποφάσεων του Συμβουλίου. Βεβαίω. Θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας στηρίξει και εμείς ευχαρίστως να σας ενημερώνουμε σε κάθε στάδιο των ενεργειών μας. Ευχαριστούμε κύριε Κωσικού, ευχαριστούμε και για την ε, καλή σας πρόθεση να μας ενημερώνετε. Για να δούμε τώρα, ε, έχουν ζητήσει ένα σωρό Το λόγο πρώτα η Ιουδίθ Μέρκες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κωσικού που μας εξηγήσατε την εταιρική σχέση για τις πρώτες ύλες, ε, τις που ανακοινώθηκε ήδη πριν ε, δύο χρόνια. Και στο πρόγραμμα Horizon 2020 βλέπουμε ότι ε, προβλέπεται ένα σχέδιο, ένα κέντρο καινοτομίας και γνώσης για τις τις πρώτες ύλες. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς θα γίνει η μετατροπή αυτό σε κέντρο καινοτομίας η προσαρμογή δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας σε ένα κέντρο γνώσης και καινοτομίας για τις πρώτες Και όταν αναφέρατε το Συμβούλιο, αλλά πότε θα επανέλθετε στο Κοινοβούλιο για να μας ενημερώσετε σχετικά με τα πρώτα αποτελέσματα ε, του EIP. Εγώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια από τις μου, διότι ε, να επενέσω και εσάς και τον Επίτροπο Ταγιάννη σχετικά με την διαθεσιμότητα πρώτων υλών και ιδιαίτερα των σπάνιων γεών. Το... Αναφερθήκατε στο θέμα της υποκατάστασης, αλλά Νομίζω ότι το βήμα πριν την υποκατάσταση είναι η αποτελεσματικότητα. Να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια αγορά για χρησιμοποιημένα, για χρησιμοποιημένες πρωτεσίλες και και προωθούνται διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα και όχι τόσο πολύ ε, διάφορα, διάφορες τεχνολογίες. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες ε, για την υποκατάσταση. Νομίζω όμως ότι το να προωθήσουμε και διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα ε, θα ήταν χρήσιμο. Θα μπορούσαμε να έχουμε ε, μια εταιρεία leasing ώστε τα προϊόντα να επανέρχονται στον παραγωγό για να μπορεί να τα ανακυκλώσει. Και τέλος, μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε Ποιο κομμάτι αυτών που μας είπατε προβλέπετε ε, για εντός της Ευρώπης και ποιο κομμάτι για χρήση εκτός της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ή τρεις παρατηρήσεις προτού να ξαναδώσω το λόγο στον ε, ομιλητή για να απαντήσει. Ο κύριο ε, Μπιτικόφερ, ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Κουζικού για την παρουσίασή του και να τον ε, συγχαρώ όχι μόνο για τις εξηγήσεις που μας έδωσε, αλλά και για την αφοσίωσή του και για την στρατηγική που ακολουθεί η Γενική του Διεύθυνση στον τομέα αυτών. Να τον συγχαρώ και για την ολοκληρωμένη προσέγγιση και ιδιαίτερα για την επιμονή σας, το πείσμα σας στην επιδίωξη των στόχων αυτών παρά, όλους του, παρά όλα τα εμπόδια που είδαμε, ιδιαίτερα σε κάποια κράτη-μέλη. Να σας πω ότι κάπως με δυσαρεστεί, για να το πω διπλωματικά, ότι η Δανέζικη Προεδρία δεν έχει βρει τρόπο να δώσει πράσινο φως ε, για αυτό το EIP ε, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ε, της χρονιάς. Εάν λίγο τους ενδιέφερε να προωθήσουν αυτό το θεματολόγιο το οποίο πιστεύω ότι είναι κεντρικό για την ε, μελλοντική ε, ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ε, καθώς και για κάποιους περιβαλλοντικούς στόχους που πάντα προέβαλαν μπορεί να ήθελα να προωθήσουν το θέμα αυτό περισσότερο. Επικροτώ τη βούληση της Επιτροπής να προοδεύσει και να μην περιμένει το Δεκέμβριο για να ε, κάνει τα απαραίτητα βήματα. Μία παρατήρηση θέλω να κάνω, διότι κύριε Κοζικού αναφερθήκατε στην έκθεση που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο. Στην έκθεση αυτή το Κοινοβούλιο ρωτά επίσης τον ε, ε, Επίτροπο και Αντιπρόεδρο Ταγιάννη ζητά από τον Επίτροπο Ταγιάννη να εκδίδει ετήσια έκθεση σχετικά με την ε, πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της πολιτικής για τις πρώτες ύλες. Από ό,τι γνωρίζω εγώ, το σχέδιο είναι να εκδοθεί μια τέτοια έκθεση ε, στο τέλος αυτής της χρονιάς ε, που να μπορεί να ενσωματώνει και τις εμπειρίες όσον αφορά το EIP. Εάν έχει αναβληθεί η επίσημη απόφαση για το EIP για το Δεκέμβριο, εγώ σας ζητώ να μην αναβάλλετε και την έκθεση. Σας ζητώ την πρώτη τέτοια έκθεση που μας υποσχέθηκε ο Αντιπρόεδρος να την υποβάλλετε εντός του έτους. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που στο πλαίσιο του ε, Horizon 2020 έχει δοθεί ένα δισεκατομμύριο ευρώ για θέματα πολιτικής των πρώτων υλών. Νομίζω ότι ε, αυτό είναι πολύ σωστό. Να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη δουλειά που κάνετε. Νομίζω όμως ότι όλοι θα πρέπει να σημειώσουμε το γεγονός ότι ε, δεν μπορούμε να αναβάλουμε το θέμα αυτό. Είναι σημαντική η δουλειά αυτή και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε όλοι μεταξύ μας και νομίζω ότι ήταν καλή η συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν στο θέμα αυτό και θα πρέπει να επιδιώξουμε πιο ισχυρά επιχειρήματα απέναντι στα κράτη-μέλη ε, ώστε να μας βοηθήσουν να μας βοηθήσουν να σπρώξουμε το όχημα αυτό προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε το συνάδελφο και τον συνάδελφο Σπριτζίνα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία. Ως γεωλόγος γνωρίζω, αντιλαμβάνομαι τι κάνετε και είναι εξαιρετικά χρήσιμος για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι η εξάρτησή μας από τις πρώτες ύλες, παρά το γεγονός ότι θαρρύνουμε την αστική εξόρυξη, την ανακύκλωση. Είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε περισσότερες προτεσίλες για το μέλλον της Ευρώπης. Η ερώτησή μου δεν θα είναι πολύ διπλωματική ίσως. Μιλούσα με την γεωλογική υπηρεσία στην Τσεχική Δημοκρατία διότι είναι αρκετά εξειδικευμένοι και τους ενθαρρύνω μερικές φορές να εμπλακούν σε, αυτές τις, ε, σε αυτή την πρωτοβουλία και μου είπαν ε, ε, αυτό είναι λίγο εδώ είμαστε ένα κλαμπ αρχαιοτέρων δεν μπορούμε να μάλλον όχι εδώ πρόκειται για ένα τομέα αρχαιοτέρων δεν μπορούμε εμείς να μπούμε σε αυτό το σύλλογο και μετά τους ρώτησα ποιο είναι το μέλλον του ΚΙΚ. Μου είπαν θα είναι οι σκανδιναβικές χώρες. Δεν ξέρω αν αυτές οι πληροφορίες είναι σωστές, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια γεωγραφική ισορροπία. Μιλάμε για κοινό ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο. Δεν θα ήταν κακό να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση σας συγχαίρω για αυτή την πρωτοβουλία και είναι πραγματικά αναγκαία για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Εάν συμφωνείτε μπορούμε να συνεχίσουμε για την επόμενη διάσταση. Συνεχίζουμε με τις δύο τελευταίες ομιλίες. Έτσι μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα το χρόνο και στο τέλος θα μπορέσετε να απαντήσετε σε όλους. Ο συνάδελφος Γκύρε και ο συνάδελφος Ρουπίκ και μετά δεν έχω άλλες ομιλίες. Ε, κύριε Γκύρε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε σε πολλές ομάδες επιφορτισμένες με τις πρώτες ύλης. Εγώ θεωρώ ότι η Λύπη ίσως η πιο σημαντική ομάδα λείπει μια ομάδα που θα μπορούσε να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιήσει αυτές τις πρώτες ύλες. δηλαδή μια ομάδα που ασχολείται με την χρήση αυτών των πρώτων υλών διότι αυτή η χρήση ουσιαστικά δημιουργεί τις βάσεις για τα ακόλουθα εκεί επικεντρώνεται ουσιαστικά η καινοτομία εκεί μιλάμε για την καινοτομία και πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα μπορεί να επιτευχθεί η μεγαλύτερη πρόοδο. σα δώσω ένα παράδειγμα. Η Ευρώπη είναι τεράστιος παραγωγός αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα, όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, ε, έχουν το αμάξωμα, 7 χρόνια εγγύσεις για ορισμένα μοντέλα ή και παραπάνω, αλλά έχουμε όλο και λιγότερο ε, καιρό για το αμάξωμα, όλο και λιγότερο και ψάχνουμε εναλλακτικέ λύσεις, ε, όπως για παράδειγμα το αλουμίνιο, το θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι για εργοστασιακές παραγωγές σε ευρωπαϊκή κλίμακα θα ήταν ωφέλιμο να αναλύσουμε από άποψη ε, χρήσης ουσιαστικά των πρώτων υλών και αφού γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τι μας λείπει, ποια υλικά μας λείπουν, ποια υλικά θα υποχρεωθούμε να εισάγουμε. Θεωρώ ότι δυστυχώς η προσέγγιση που υιοθετείται είναι η αντίστροφη. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την άλλη ε, άκρη. Ευχαριστώ. Η τελευταία ομιλία ο κύριος Ρούμπι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε επικροτώ την πρωτοβουλία. Είναι μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση αυτή που αναζητούμε εδώ στην Ευρώπη και οι πόροι της Ευρώπης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Γι' αυτό σκεφτόμαστε τις υποδομές που χρειαζόμαστε για τις πρώτες ύλε. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Αυτή τη στιγμή στο ε, κοινό ερευνητικό κέντρο στο Μιλάνο υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο εξετάζει διάφορα θέματα βιοπικιλότητας, ε, των ε, ε, οδών μεταφορών. Θα πρέπει να εξετάσουμε και τι εκτάσεις θα χρειαστούν μακροπρόθεσμα θα πρέπει να γίνει ευρωπαϊκός συντονισμός. Σημαντικό είναι να κοιτάξουμε τις περιβαλλοντικές πτυχές ε, με επιστημονική βάση και να εκπονήσουμε επιστημονικές συμβουλές ώστε να μην είμαστε αυτομάτως ε, κατά οποιοδήποτε νέου ε, προγράμματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπιτικόφερ, διότι αυτός παρουσίασε τον συλλογισμό ότι οι προτάσεις ε, των ε, περιβαλλοντολόγων θα πρέπει να ε, εξετάζονται όσον αφορά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων. Όταν μας λέμε ότι ναι, αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να το πραγματοποιήσετε, ενώ ίσως είναι καλύτερα να περιμένετε με το άλλο. Είναι Φυσικά σημαντικό και το θέμα στον ορίζον 2020 να εξετάσουμε ποια, σε ποιους τομείς μπορούμε να δώσουμε βάρος και και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας να κοιτάξουμε και ε, τι προγράμματα εκπαίδευσης είναι δυνατόν να γίνουν και πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της φορολογίας, ε, των μεταφορών σε μεγάλες αποστάσεις. Ε, να εξετάσουμε την φορολογία που μπορεί να επιβληθεί ώστε ενδεχομένω οι πρώτε ύλε που πρέπει να μεταφερθούν ε, σε μεγάλες αποστάσεις ε, να πληρώνουν 2-3% περισσότερο ΦΠΑ. ώστε από οικονομική πλευρά ε, να δώσουμε προτεραιότητα στις πρώτε ύλε που βρίσκονται πιο κοντά. Ευχαριστώ πολλές ερωτήσεις σε αυτέ τι πέντε ομιλίε. Παρακαλώ τώρα να δώσετε τι απαντήσει. Σα ευχαριστώ πολύ ευρείες αυτές οι ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να μην ξεχάσω τίποτα. Η σχέση μεταξύ του IP και του KIC. Πιστεύω ότι το σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι είναι συμπληρωματικά. Δεν υποκαθιστά το ένα το άλλο. Το EIP είναι συνεργασία για την καινοτομία, το KIC είναι για τις δεξιότητες καινοτομίας. Όταν μιλάμε λοιπόν για EIP είτε για KIC θα ισχύει για ό,τι και αν συζητάμε δεν αντικαθιστά το ένα το άλλο. Έχουν έτσι σχεδιαστεί από την αρχή, ώστε να είναι συμπληρωματικά. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τη διάρκεια του EIP. Δεν έχουμε προβλέψει κάποια λήξη. Είναι σαφές ότι συνδέεται στενά από απόψεις πρακτικής με το Horizon 2020. Επίσης είναι σαφές ότι το ζήτημα των πρώτων υλών δεν θα πάψει να υπάρχει αύριο θα υπάρχει για αρκετό καιρό. Ακόμη και αν δουλέψουμε σκληρά, πρόκειται για ένα ζήτημα που θα διαρκέσει για πολλέ δεκαετίε. Όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, η ίδια η γνωμοδότηση αποτελεί απάντηση αυτό, τον όσων ζητήσαμε στο ψήφισμα. Υλοποιούμε αυτά που μας ζήτησε το Κοινοβούλιο να πράξουμε και το Σεπτέμβριο μας ζητήσατε να ξεκινήσουμε μια σύμπραξη καινοτομία έγινε το Φεβρουάριο και εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε προνομιακή απόδοση, τεχνολογία, τεχνολογία την κατάσταση. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Εάν σας έδωσα μια τέτοια εντύπωση, αυτό οφείλεται στο ότι ήταν πολύ σύντομη η παρουσίασή μου Πιστεύω ωστόσο ότι προλαβαίνω να πω ότι δεν είναι μόνο τεχνολογία και το ανέφερα και στις πέντε ομάδες εργασίας ότι οι δύο ε, εστιάζονται στην τεχνολογία και δύο όχι. Είναι σαφές ότι πέραν των τεχνολογικών λύσεων που θα χρειαστεί να αναπτύξουμε υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσουμε όπως οι δημόσιες προμήθειες, η τυποποίηση και οι πολιτικές τυποποίησεις και επιστοποίησες, Το ανέφερα και στην παρουσίασή μου νομίζω. Η σχέση με το τι, μεταξύ του τι θα γίνει και του διεθνού στοιχείου. Το διεθνή στοιχείο είναι σημαντικό όταν συζητάμε ερευνητικές προτεραιότητες, ερευνητικά προγράμματα σε δοκιμαστική βάση. Έχουμε ξεκινήσει ήδη με την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σαφές ότι πρέπει να αυξηθεί η ροή πληροφοριών και ο διάλογος τόσο για τεχνολογία όσο και για άλλα θέματα. Όταν αναπτύσσουμε πολιτικές πρέπει να δούμε μαζί με τους συνεργάτες μας, με τους εταίρους μας αν έχουν καλύτερες ε, απαντήσεις για τις ερωτήσεις που θέτουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν ε, ε, θεωρούμε ότι γνωρίζουμε την απόλυτη αλήθεια. Κύριε Μινκόφερ, ευχαριστώ για τα συγχαρητηριά σας και για το, την ενθάρρυνση που προσφέρετε. Όσον αφορά τις τακτικές αναφορές και εκθέσεις, ε, είναι σαφές ότι θέλουμε να έχουμε τακτικές εκθέσεις έχουμε επιδείξει την πρόθεσή μας ε, ότι οποτεδήποτε το Κοινοβούλιο θέλει να ενημερωθεί δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Και ο κ. Μπουζίνα ανέφερε την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Την ίδια ανησυχία έχουμε και εμείς δεν θα βρούμε θαυματουργές λύσεις για ένα τομέα που θα λύσει ολόκληρο πρόβλημα. Πρέπει να κοιτάξουμε όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Τα σχόλιά σας ε, τα ανέφερα στην υπηρεσία μου. Δεν υπάρχει κάτι, ε, κάποιος και κάποια ανησυχία. Θα πρέπει να δούμε την κατάσταση με τους αρμόδιους συναδέλφους. Ο κύριος Γκέρακ ανέφερε την ανάγκη για να επικεντρωθούμε και στη χρήση των πρώτων υλών. Έχουμε κάνει κάποια πράγματα σε αυτό το τομέα. Εντοπίσαμε τον κατάλογο των κρίσιμων πρώτων υλών. Θα ξαναμελετήσουμε αυτόν τον κατάλογο από φέτος, ώστε του χρόνου το 2013 να δούμε κατά πόσο θα συνεχίσει να ισχύει. Επίσης, Ξεκινήσαμε μια μελέτη για τις ροές πρώτων υλών. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Οι αλυσίδες αξίας είναι εξαιρετικά πολύπλοκες. Το να γνωρίζει κανείς ε, που γίνεται η επεξεργασία και που καταλήγει μια πρώτη ύλη είναι τρομακτικά περίπλοκο, αλλά έχουμε συνείδηση της ανάγκης αυτής. Κύριε Ρίμπικ, αναφέρετε τις υποδομές για τις πρώτες ύλες. Αληθεύει αποτελεί κομμάτι του δεύτερου πυλώνα της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες. Έχουμε ήδη δουλέψει για το Natura 2020 τις ε, δραστηριότητες εξόρυξης αλλά το Natura 2020 δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε εξορυκτικές δραστηριότητες κοντά στο Natura 2000 τηρώντας φυσικά τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις η δική σας χώρα, μάλιστα, καταγωγής είναι πολύ δραστήρια σε αυτές τις πρακτικές και βοηθάει και μας υποστηρίζει πάρα πολύ στο να προωθήσουμε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, τη χρήση γης, το χωροτεξικό σχεδιασμό και ούτω καθεξής. Το ίδιο θα ισχύσει και για άλλους τομείς, όπως τη θαλάσσια πολιτική, γιατί και εκεί χρειάζεται να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας όσον αφορά τις προϋποθέσεις περιβάλλοντος για να έχουμε πρόσβαση στις αναγκαίες πρώτες ύλε. Όσον αφορά τώρα τη φορολόγηση των εταιριών δεν θα σχολιάσω, αλλά φαντάζομαι ότι αφορά περισσότερα τις πολιτικές ενεργειακής φορολόγησης παρά τον τομέα των πρώτων υλών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και για τις απαντήσεις σας. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι όπως συνήθως μετά από αυτή τη συζήτηση και την παρουσίαση της πρότασης ε, θα λάβετε μια επιστολή από την πρόεδρο της Επιτροπής μας που θα προσπογραφεί από τους συντονιστές και με αυτή την επιστολή θα μπορούσατε να λάβουμε τυχόν υποδείξεις, προτάσεις που δεν υπήρχαν στις προτάσεις που ακούσαμε και που δεν είχαν ε, αναδειχθεί πλήρω. Ε, παρακαλώ λοιπόν του συναδέλφου να μα στείλουν τι παρατηρήσει του, ώστε η επιστολή αυτή να αποτελεί το αποκύμα αυτή τη ε, ενδιαφέρουσα συζήτηση για την οποία και πάλι σα ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Αποχαιρετούμε τον κύριο Κοτσίγκου. Ασφάλεια των δραστηριοτήτων ότρε εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου ανοιχτή θαλάσση. Εισηγητή κ. Μπελέτ. Υπενθυμίζω ότι ο χρόνος που είχε προβλεφθεί ήταν περίπου 60 λεπτά και τώρα αναγκαστικά τον μειώνουμε σε 40. Έτσι λοιπόν θα μειώσουμε και τους δικούς μας χρόνους διότι είναι το τελευταίο σημείο και φυσικά υποφέρει από όλες τις ισορρευμένες καθυστερήσεις. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο στην Μπελέτη. Ε, <clears throat> Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Μπέλετ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε την ευκαιρία τώρα να αρχίσουμε τη συζήτηση για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Όπως γνωρίζετε, άργησε το θέμα αυτό να προωθηθεί γιατί καθυστέρησαν να το διεκπαιριώσουν οι συναρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Πρώτα πρώτα να σας πω μερικά πράγματα όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο γιατί έχουμε βέβαια τη συνάντηση με τους εισηγητές των άλλων επιτροπών. Έγινε αυτό σήμερα το πρωί στις 9 Οκτωβρίου η ΕΝΒΗ που έχει κάποιες αμπουλιστικές αρμοδιότητες για το θέμα έχουμε κάποιες κοινέ με την ΕΝΒΗ και επίσης αυτό ισχύει και για την Συναρμοδιονομική Επιτροπή Παραμένουμε όμω ε, η κυρίω αρμόδια επιτροπή. Όμως η ΕΝΒΗ έχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο ξεπερνά αυτό το οποίο εμείς καταρχήν ορίσαμε σε σχέση και με την τελική ψηφορία. Άρα ήρθαμε σε επαφή με την ΕΝΒΗ αυτό το θέμα. Ε, αυτοί διστρόπησαν λίγο, είναι όμω πάρα πολύ σημαντικό. Το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται βέβαια να προωθεί το ζήτημα και επομένω και αυτό είναι και ο στόχο ημών αλλά και όλων των καταναλωτών που να μπορέσουμε το συντομότερο δυνατόν να πετύχουμε συμφωνία και να υπάρξει το καινούριο πλαίσιο. Οπότε το συντομότερο δυνατόν ελπίζουμε να λυθεί το πρόβλημα μετά τη συμφωνία με την Ένδια. Και έτσι να έχουμε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Δεν χρειάζεται να σας επαναλάβω το πώς τι έγινε πριν από δύο χρόνια με το ατύχημα στον κόλπο του Μεξικού. Είχαμε 11 νεκρούς, 5 εκατομμύρια περίπου αργού πετρελαίου χύθηκαν στη θάλασσα ε, και όλοι θα θυμάστε τα γεγονότα καλά. Αμέσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την ε, μελέτη των επιπτώσεων κατέληξαν στο ότι θα πρέπει να λυθούν ενέργειες και για την Ευρώπη. Έτσι ξεκίνησε αυτό το σχέδιο κανονισμού, το οποίο τώρα βρίσκεται στις τραπέζες. Βέβαια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας δεν φνηδιάζονται από όλα αυτά μια που ήδη στο παρελθόν ήμασταν έτοιμοι, είχαμε αξιόλογη προετοιμασία, είχαμε και τη σχετική έκθεση, το σχετικό ψήφισμα. Ε, της κυρίας Φόρτ ε, πέρσι, πέρσι με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε. Οπότε και το Κοινοβούλιο είχε ξεκάθαρη άποψη για το θέμα τώρα. Θα πρέπει να σας ε, υπενθυμίσω ότι το Συμβούλιο ήδη έχει προχωρήσει το θέμα. Το είπαμε και στην αρχή, χάθηκε λίγος χρόνος. Το Συμβούλιο όμως δεν περίμενε. Η πρόοδος συνεχίστηκε και η ομάδα εργασία του Κοινοβουλίου το συζήτησε και το ξανασυζήτησε. Η ΔΕ, Δανέζικη Προεδρία, πριν ολοκληρωθεί, θα προχωρήσει σε σχετική έκθεση, σχετική δημοσίευση, το οποίο θα γίνει περί τις 15 Ιουνίου. Και για το δεύτερο ή της, ε, του έτους πρόκειται να προχωρήσουμε στον τριμερή διάλογο. Τώρα, τι γίνεται όσον αφορά αυτό το σχέδιο κανονισμού. Σήμερα, συνάδελφε, πάνω από 90% του πετρελαίου και πάνω από 60% του φυσικού αερίου που παράγεται στην ε, Ένωση ε, βγαίνει από την θάλασσα. Δηλαδή, έχουμε πάνω από Βέβαια, πάρα, πάρα πολλέ τέλο πάντων ε, τέτοιε υπεράκτητε εγκαταστάσει εξόριξη στην Ευρώπη. Κυρίω στη Βόρεια Θάλασσα. Βασίλειο, Νορβηγία. Παντού όμως όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γίνεται παραγωγή. Δανία, κάτω χώρες, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Μάλτα, Κύπρο, 13 κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει σε τέτοιου είδου αδειοδοτήσει εξόριξη. Ε, υπάρχει. Επομένω, αυτό γίνεται παντού. Δεν γίνεται μόνο στην Μαύρη Θάλασσα. Παντού και στην Μεσόγειο. Και επομένω. Και κατά τον τρόπο έχουμε διάφορες, ε, διάφορους κανόνες σε σχέση με τα πρότυπα, τις παραγωγές και λοιπά και γι' αυτό και ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η προηγουμένη νομοθεσία δεν εκάλυπτε όλες αυτές τις πτυχές. Οπότε, για να δούμε τώρα. Ποια είναι τα βασικά σημεία της πρότασης. Είναι αρκετά τεχνοκρατική, εγώ θα περιοριστώ στις βασικές γραμμές. Ο στόχος είναι πρώτα πρώτα να προλάβουμε μια άλλη τραγωδία, να μην γίνει. Και επίσης να δούμε το πώς θα είμαστε έτοιμοι αν κάτι γίνει. Πρώτα πρώτα, όσον αφορά την διαδικασία διοδότησης, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι μόνο όσοι έχουν τα προσόντα, τις ικανότητες, τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν διαδικασίες χωρίς κίνδυνα μόνο αυτοί θα έχουν την άδεια για την εξόριξη. Άρα, κανείς αν θέλει να μπλεχτεί σε αυτό θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα προσόντα και δυνατότητες. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει να γίνεται ανεξάρτητη επαλήθευση η ασφάλεια στις εγκαταστάσεις θα διαπιστώνεται επομένως, θα επαληθεύεται από κάποια αρχή ανεξάρτητη. Τρίτον, κάποιος προγραμματισμός του κατεπίγουσης φύσεως θεμάτων θα είναι υποχρεωτικός και πάρα πολύ σημαντικός. Επίσης θα πρέπει ανεξάρτητες, ε, ανεξάρτητη αρχή, ανεξάρτητη φορείς θα πρέπει να διαπιστώνουν την ασφάλεια και για το περιβάλλον και επίσης κάτι άλλο ότι είναι η διατάξη σε σχέση με την ευθύνη. Οι εταιρείε που ασχολούνται με φυσικό αέριο και πετρέλαιο θα έχουν πλήρη, πλήρη, πλήρη ευθύνη σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό για κάθε βλάβη προ το περιβάλλον που δημιουργήθηκε από την ε, παραγωγή, για το περιβάλλον, το φυσικό, τα, τα, τα, θαλάσσια, θάλασσα τέλο πάντων. Σε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο τώρα. Ποια είναι τα πιο σημαντικά σημεία του κανονισμού. Το θέμα είναι που συζητείτε το κατά πόσο θα πρέπει να γίνει κανονισμός ή να γίνει οδηγία. Έχει προτείνει κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεώρησε ότι αυτό είναι το νομικό μέσο που προσφέρεται γιατί έτσι θα έχουμε θεμητούς ως ανταγωνισμού. Θα έχουμε επίσης ομοιόμορφη προσέγγιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω, ξέρουμε ότι η οδηγία απαιτεί μεταφράσει στο ιστορικό δίκαιο. Οπότε εκεί έχουμε διαφοροποιημένα αποτελέσματα ανάλογα με το κράτος μέλος. Πολλοί επίσης από τους εμπλεκόμενους σε επίπεδο αλλά και κάποιες εθνικές αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο θεωρούν ότι ο κανονισμός θα δημιουργήσει κάποια αβεβαιότητα σε σχέση με το νομικό πλαίσιο. Επίσης, θα πρέπει να καταργηθεί ό,τι πλαίσιο ε, ότι, ότι νομικό πλαίσιο ισχύει σε κάποια σε χώρες μέλη, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε μία ομοιόμορφη αντιμετώπιση να ευθυγραμμιστούμε. Αυτό όμως θα πάρει χρόνο. Και ίσως αυτό είναι ει βάρο τη ασφάλειας. Πάντως θα πρέπει οπωσδήποτε να καταβληθεί προσπάθεια τέτοιων ε, προσαρμογών σε νομικό επίπεδο. Κάτι άλλο επίσης ε, σημαντικό είναι οι παρατηρήσει των εμπλεκομένων όσον αφορά την μελέτη των επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. σας υπενθυμίζω κάτι το οποίο ίσως όλοι το γνωρίζετε ότι στο μέλλον η παραγωγή πρόκειται να γίνεται η εξόριξη τέλο πάντων σε βαθύτερα ύδατα. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο. Και να ληφθεί επίση υπόψη ότι αυτά θα γίνονται και σε πολύ μακρινά σημεία της υδρογείου όπως στην Αρκτική. Οπότε εκεί θα αντιμετωπίσουμε κινδύνου και προκλήσει καινούργιε. Κύριε Πρόεδρε, περιορίστηκα στα πιο βασικά σημεία. Αυτά που αφορούν την ε, Ήτρε. Υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία αφορούν ή αφορούν μόνο ή και την Επιτροπή Περιβάλλοντος και την Νομική Επιτροπή. Όπως είπαμε, ε, Φερρυπίν, το θέμα της ευθύνης τους καταγγέλλοντες ε, και την αντιμετώπιση του όσον αφορά του καταγγέλλοντε ε, εργαζομένους. Πριν από λίγες εβδομάδε είχαμε σε μια πλατφόρμα τη Total κοντά στο Αμπερντίν άλλο ένα ατύχημα και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει τέλεια εγκατάσταση που να μην ε, έχει πιθανότητες ατυχημάτων. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, πρέπει να τα κάνουμε καλύτερα και επίσης θα πρέπει να γίνει εις βάθος έρευνα του τι πήγε στραβά. Και να δούμε επομένως τι βελτιώσεις θα κάνουμε και τέτοιους έρευνε βέβαια προβλέπονται και στον συζητούμενο οργανισμό. Ευχαριστώ να ακούσω τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα επίση να διαβεβαιώσω το συνάδελφο εισηγητή και όλους τους συναδέλφους ότι θα ξανά έχουμε χρόνο για συζήτηση όταν θα παρουσιαστεί το σχέδιο γνωμοδότηση 11 και 12 Ιουλίου. Δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα λοιπόν σήμερα. Τέσσερι σκιώδει και λοιπέ ομιλίε, πολύ περιορισμένη χρόνη, παρακαλώ και για τους σκιώδει, όχι πάνω από τρία λεπτά, μπορείτε να το δείτε. Και στον οθονή το λόγο είχε ο Συνάδελφο Σκίνερ, πρώτο σκιώδη των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον Ήβο για την εισαγωγή του. μας ε, θυμίζουν όλα αυτά ε, διαμαρτυρίες από ε, τον βιομηχανικό τομέα εδώ και κάποια χρόνια ότι δεν επιτρέπεται να λιμνάζουν τα πράγματα και ότι πρέπει να υπάρχουν πρότυπα για την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και θα επανέλθω σε αυτό στις μελλοντικέ συζητήσεις που μας θύμισε η Πρόεδρος ότι θα έχουμε. Νομίζω ότι οι βέλτισες πρακτικές ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε και να χρησιμοποιούμε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, το θέμα αν θα πρέπει να είναι οδηγία ή κανονισμός το θέμα της εξόριξης πετρελαίου σε βαθέα ύδατα είναι λίγο αδιάφορο τη στιγμή που λιγότερο από το μισό των κρατών μελών συμμετέχει σε τέτοιες δραστηριότητες. Ξέρω ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ε, έχουν ε, μιλήσει μαζί μου για σημαντικά θέματα τα οποία αναφέρατε εσείς ήδη, όπως είναι οι, ε, οι υπεράκτιες εξορίξεις πετρελαίου offshore. Ξέρω ότι θα το ακούσετε αυτό και από άλλους εισηγητές. Σημαντικό είναι να υπάρχει η διαφοροποίηση των ε, του όφελους ε, της εξόριξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Γι' αυτό χαίρομαι που ε, η Κομισιόν έχει θέσει μορατόριο για το θέμα αυτό, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να ενεργήσουμε καθόλου. Αλλά θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε προβλήματα όπως το ατύχημα που είχαμε με την διαρροή αερίου ε, πριν ε, λίγες μέρες ε, να μην μας εμποδίσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας στον τομέα αυτών. Να κλείσω εδώ να... Πω μόνο ότι ε, οι εξορίξεις πετρελαίου ε, στις ακτές της Ευρώπης ε, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που γίνονται στο Μεξικό. Εμείς έχουμε θέσει κάποια όρια, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα όρια τα δικά μας απέχουν πάρα πολύ από τα όρια του Μεξικού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Σκίνερ για τα όσα είπε και που τήρησε το χρόνο. Ευχαριστούμε φιόν Ευχαριστώ. Ε, να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπέλετ ε, για την έκθεσή του. Θα ήθελα να αναφέρω λίγα θέματα λόγω της πίεσης του χρόνου. Καταρχήν έχουμε ε, το θέμα κανονισμού ή οδηγίας. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό ότι αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα επαχθές για χώρες ε, που ήδη ε, έχουν ε, ένα καθιερωμένο καθεστώς εάν πρέπει να ανατρέψουν όλο τους το σύστημα. Ή θα πρέπει να έχουμε οδηγία τελικά πιστεύω ή θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στο Συμβούλιο που είναι μπροστά από μας στις συζητήσεις αυτές όπου ε, φαίνεται να ε, ε, διαφαίνεται κάποια δυνατότητα, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να καταλήξουμε να σπαταλάμε πολύτιμο χρόνο και δυναμικό προσπαθώντας να επανεφεύρουμε το τροχό τη στιγμή που ήδη έχουμε πολύ καλά παραδείγματα νομοθεσία στη διάθεσή μα. Δεύτερον, θα ήθελα να επικροτήσω την απόφαση τη Κομισιόν ε, να δημιουργήσει την ε, ομάδα για τι ε, υπερακτίε εξορίξει φέτο το καλοκαίρι, διότι έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε χρησιμοποιώντα την εθνική εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει. Όσον αφορά την διασφάλιση τη συμμόρφωση από τα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, αν ε, λοιπόν ε, έχουμε οδηγία με πιο ελεύθερο καθεστώς για τα κράτη-μέλη, σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση και δίδεται έτσι η δυνατότητα να διασφαλίσουμε την συμμόρφωση με λίγο διαφορετικό τρόπο, αντί να πρέπει να ε, διαβρύνουμε την εντολή της ε, ΕΜΣΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, συζητήθηκε και στο πλαίσιο της έκθεσης Ford. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε ένα σύστημα ανεξάρτητο και όχι ιδιαίτερα επαχθές. Είναι ευάλωτο τομέα και δύσκολο ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερα καθεστώ ε, για τις δραστηριότητε που αφορούν το πετρέλαιο και το αέριο. πόσο μάλλον που ο σχεδιασμός ε, αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι κάτι το οποίο Ε, είναι πιο δύσκολο ε, στα βόρεια ύδατα από ότι στα ε, πιο νότια και θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στον τομέα της ε, κατανομής νερού. Θα ήθελα πολύ να δω ε, τα σχέδια ε, αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσουμε την διαφάνεια. Σημαντικό είναι να έχουμε μηχανισμούς παρόμοιους με αυτούς της του τομέα αερομεταφορών. Δηλαδή, αν κάτι πάει στραβά, το σύνολο του τομέα να μαθαίνει από αυτό και να διορθώνει την κατάσταση. Και επίσης, ε, το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας μπορεί να επιτευχθεί από ευρωπαϊκές εταιρείες που να εργάζονται εκτός των υδάτων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι δύσκολος τομέας, αλλά μπορεί να διασφαλιστεί αυτό. Οι ενωσιακές επιχειρήσεις ε, δηλαδή να ε, τηρούν τα ίδια πρότυπα σε όλο τον κόσμο και θα πρέπει να είναι δυνατόν να προσφύγει κανείς σε ευρωπαϊκά δικαστήρια σε περίπτωση παραβάσεων όπως κάνουμε και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο της ε, οδηγίας για την διαφάνεια. Ζητάμε από τις ευρωπαϊκές εταιρείες να μας ε, δηλώνουν τι πληρώνουν ε, οπουδήποτε στον κόσμο. Με παράλληλο τρόπο μπορούμε να απαιτήσουμε από τις ευρωπαϊκές εταιρείες να πληρούν τα ίδια πρότυπα ασφαλείας σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Φιονόλ, Τον λόγο έχει η κυρία Ναβαζή. Άνευ μικροφώνου η ομιλήτρια. Ευχαριστώ τον εισηγητή όσον αφορά το ζήτημα του κανονισμού της οδηγίας. Εγώ έμαθα ότι το Συμβούλιο αντιτίθεται από τις 25 Μαΐου στο γεγονός ότι υπάρχει κανονισμός. Όπως αναφέρατε, εάν συντάξουμε μια οδηγία θα πάρει χρόνο και μετά θα υπάρχει διάκριση μεταξύ των χωρών όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας. Εμείς ωστόσο θέλουμε να κάνουμε γρήγορα και θέλουμε να αφορά όλες τις χώρες ε, να τους επιβάλλει υψηλά πρότυπα ασφαλείας. Και επίσης το ατύχημα δεν πρόκειται να περιμένει. Εάν ο κανονισμό αφορά όλε τι χώρε τόσο πιο λειτουργικοί θα είμαστε. Είμαι λοιπόν υπέρ του κανονισμού. Το δεύτερο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι υπάρχει ανάγκη για ευρωπαϊκό οργανισμό, ευρωπαϊκή υπηρεσία. Πώς επεκτείνουμε τα προνόμια της ΕΜΣΑ, συζητώντας με τους βιομηχάνους, μου λένε εμείς έχουμε τα ύψιστα πρότυπα, μόνο που υπάρχουν πολλές εταιρείε και πρέπει να υπάρχει ένας ανεξάρτητο οργανισμός, ο οποίος να μπορεί να ελέγχει ε, κατά πόσο αληθεύουν όσα λένε η πετρελαιοπαραγωγή και οι βιομηχανή. Επίση, πρέπει να εξετασούμε τους κίνδυνους ε, διένεξης συμφερόντων μεταξύ πετρελαιοπαραγωγών και κρατών μελών. Στη συνέχεια θα πρέπει επίσης να μαθαίνουμε και κάποιο σχολιασμό από τις διάφορες εμπειρίες. Όταν γίνονται ατυχήματα, αυτό που είναι ενδιαφέρον να αναλύουμε αυτά τα ατυχήματα και να τα κοινοποιούμε σε όλους ώστε να μπορούμε να βρούμε μια λύση σε περίπτωση ατυχήματος και να μπορούμε να προβούμε σε προληπτικές ενέργειες για άλλα ατυχήματα. Αυτό θα είναι ο ρόλος αυτού του οργανισμού για αυτό το λόγο και εμείς είμαστε πιο ευνοϊκοί για τη λύση 3. Δηλαδή να υπάρχει ευθύνη των κρατών μελών σε σχέση με τους οργανισμούς και των βιομηχάνων αλλά να υπάρχουν και οι δυνατότητες επιθεώρησης και έρευνας από αυτόν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Στη συνέχεια, όσον αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις, χαίρομαι που η πρόταση της Κομισιόν για την επέκταση της οδηγίας των περιβαλλοντικών ε, ευθυνών στις πλατφόρμες offshore θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε την ευθύνη των φορέων για τυχόν περιβαλλοντικές ζημιέ και ειδικότερα όταν δρούν σε αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Βλέπετε, στη Γαλλία υπάρχει το παράδειγμα τη Ερικά που δεν είναι υπεύθυνη διότι βρίσκεται σε αυτή την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όσον αφορά την ποινικοποίηση των παραλήψεων πιστεύω ότι οι ε, μαύρες κοιλίδες θα πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη για την περικοπήση των ατυχημάτων λόγω ε, Όταν μιλάμε για τις SCP τώρα, είναι σημαντικό να μην έχουμε διπλά πρότυπα. Δηλαδή, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν τα ίδια επίπεδα, τα ίδια πρότυπα όταν δρούν στο εξωτερικό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε ευρωπαϊκά δικαστήρια σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, διότι σε ορισμένες περιοχές όπως το Δέλτα του Νίγερα για παράδειγμα, έχουμε τεράστιες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα όπως και στη Βόρεια Θάλασσα. Και το τελευταίο, απογοητεύτηκα λίγο από την προβληματική έρευνα και ανάπτυξη. Θα ήθελα οι επιχειρήσεις να έχουν την υποχρέωση να αφιερώνουν ένα μικρό ποσοστό του κύκλου εργασιών τους για την έρευνα τη πρόληψη σε περίπτωση ατυχήματο. Κοιτάξτε αυτό που έγινε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Χρειάστηκε να περιμένουν μήνες για να κατασκευάσουν αυτό το χωνί ώστε να περιορίσουν ε, τη διαρροή. Είναι απίστευτο και εδώ μιλάμε για έλλειψη πρόληψης της μελέτης επιπτώσεων είτε μιλάμε για το ίδιο το υλικό είτε για όλα τα τεχνικά μέσα που χρειάζονται για να ε, περιορίζουν την διαρροή. Λοιπόν, μας λείπει ο κύριος Φόρντ, τελευταία ομιλία σκιώδους από το, ε, της ε, κυρίας Φόρντ από το ECR. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε όλους όσους δουλέψανε τόσο σκληρά ε, αποτελούν το πετρέλαιο και το αέριο κρίσιμο κομμάτι στο μείγμα ενέργειάς μας, περιλαμβάνουν σημαντικούς κινδύνους, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλή για τους εργαζομένους και ότι θα έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Όσον αφορά αυτές τις επιπτώσεις, η εκτίμηση εκτυπώσεων, ε, ε, επιπτώσεων πιστεύω της Κομισιόν έχει ελλείψεις ε, δίνει τα ίδια κριτήρια για τα πάντα όπως και για τον κόλπο του Μεξικού και όπως το ανέφερε ο Πίτερ δεν είναι όλα υψηλής πίεσης πράγματι στην Βόρεια Θάλασσα λιγότερα από τα ε, ε, λιγότερες από τις μισές γεωτρήσεις θα παρουσίαζαν ροή σε περίπτωση που υπήρχε διαρροή αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα με τον κανονισμό σε σχέση με την οδηγία. Δεν είναι απλά το κόστος υλοποίησης, αλλά και το ζήτημα του κατά πόσο εφόσον ε, το υλοποιήσουμε αυτό ε, χάνουμε ε, ποιότητα. Ο κανονισμός θα υλοποιηθεί σε πέντε χρόνια και η οδηγία θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε δύο. Και αυτό έχει να κάνουμε με το να αλλάξουμε τι εκθέσει ασφαλεία σε κάθε εγκατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η νομοθεσία πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε να αναβαθμίσει τα πρότυπα ασφαλεία όλων και όχι να αφήσει νομικέ αβεβαιότητε. Συμφωνώ με τη Φιώνα ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι, κανονισμό, οδηγία ή σημαντική αλλαγή στη διατύπωση. Αλλά ίσω η οδηγία να είναι η ευκολότερη προσέγγιση βραχυπρόθεσμα. βραχυπροθεσμα και δεν είναι γιατί θέλουμε να ψηφίζουμε η ποιότερη νομοθεσία, αλλά καλή νομοθεσία όσον αφορά την πρόληψη. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι πρέπει να φροντίσουμε οι προϋποθέσεις ασφαλείας να μην, και οι εκθέσεις ασφαλείας να μην είναι στατικές, να εξελίσσονται με το χρόνο και να αποτελούν κομμάτι, ε, αναπόσπαστο κομμάτι της ασφάλειας. Όσον αφορά την επαλήθευση των τρίτων μερών, Υπάρχουν φορές όπου και ένας δεύτερος επαληθευτής ε, είναι χρήσιμος, άλλες φορές όχι. Για παράδειγμα σήμερα η BP έχει ε, υπευθύνου αξιολόγηση τρίτους που έρχονται και αξιολογούν τον εξοπλισμό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πότε χρειάζονται τρίτα μέρη και πότε όχι. Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν ωφέλιμο. Όταν συμβεί ατύχημα, όπως είδαμε στο Άλγκαν, Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν τα σχέδια απόκρισης, εκτακτής ανάγκης. Αυτό συνέβησε στην έργα. Σωστό σχέδιο και σωστό προσωπικό, εκπαιδευμένο σωστά, σημαίνει ότι δεν πέθαναν άνθρωποι, ότι η ρήπανση ήταν αμεληταία, ακόμη και για τους πιο ανήσυχους περιβαλλοντολόγους. Αυτό είναι πολύ καλό ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όταν συμβαίνει ένα ατύχημα μπορούμε να το ελέγξουμε. Ο εξοπλισμός κάπινγκ και περιορισμού είναι πολύ καλή εξέλιξη, πολύ καλές εξέλιξεις επίσης η ύπαρξη φρεατίων ανακούφισης, ανακουφιστικών φρεατίων ε, για τα σενάρια πιο υψηλού κινδύνου, η κοινοποίηση πληροφοριών και η εκμάθηση από τα διδάγματα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Ο GP έχει αρχίσει να μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να του βοηθήσουμε ώστε να κάνουν τα πράγματα σαφίστερα. Η ευθύνη του ρηπαίνοντο είναι πολύ σημαντική. Ο ρηπαίνον πρέπει να πληρώνει. Το πώ πληρώνει όμω και το πώ αποδεικνύει ότι έχει τα μέσα να πληρώσει είναι ένα άλλο θέμα. Εκεί πιστεύω η Επιτροπή Περιβάλλοντο δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα όταν μπαίνουμε και αρχίσουμε και συζητάμε για χρηματοοικονομικά μέσα προσπαθούν να το αναφέρουν στην ίδια πρωτοβουλία εκθεσή τους. Υπάρχει μια τεράστια αγορά ασφαλιστικών μέσων για αυτές τις δραστηριότητες και θα πρέπει να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες όλων αυτών ε, Επίσης, οι των οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης ανησυχούν για το κατά πόσο η βιομηχανία είναι έτοιμη να μπορέσει να διασφαλίσει εκ των προτέρων. Με ανησυχεί το χρονοδιάγραμμα της ΕΝΒΗ. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε λίγα δευτερόλεπτα. Οι αρχές ε, για το offshore θα λειτουργήσει μόνο εφόσον η Κομισιόν είναι έτοιμη να ακούσει αυτά που έχουν να πούν. Εάν είχε ακούσει η Κομισιόν τι θα είχαν πει πριν ε, δημοσίευση αυτόν τον κανονισμό, δεν θα είχε χρειαστεί να υποβάλουμε τόσε πολλέ τροπολογίε. Ευχαριστούμε. Τώρα σας παρακαλώ όλους να, συνεργαστείτε, όλους να συνεργαστείτε μαζί μου για τα συμπεράσματα αυτού του πρωινού. Έχουμε τρεις ακόμη ομιλίες Κομισιόν και ο εισηγητής πρέπει να κλείσει. Ζητώ λοιπόν από τον κύριο Σμίθ και Βινταλκουάδρ και Δεκαστήγιο να παραμείνετε στα δύο λεπτά παρακαλώ διότι διαφορετικά δεν θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Σμιτ. Πρόεδρε ευχαριστώ. Χαίρομαι για το πνεύμα της σημερινής συζήτησης. Χαίρο τον εισηγητή. Πολύ ισορροπημένη αξιολόγηση των πραγματών και του πιθανής έκβασης. Χαίρομαι. Ε, προερχόμενος από τη Σκοτία που το παίρνουμε όλοι τόσο σοβαρά όλα αυτά γιατί για μας εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό εθνικό θέμα. Δεν θέλουμε να μας κάνουν μαθήματα για τα πρότυπα ασφαλείας. Έχουμε, είχαμε πικρά διδάγματα ως ε, κράτος. Έχουμε κοινή φιλοδοξία. Αυτό το έχουμε συμφωνήσει. Θέλουμε να υπάρχουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για τους εργαζομένους και για το περιβάλλον. Το ζήτημα είναι ότι προς τους νομοθέτης είναι ότι αυτή η δέσμη μέτρων θα το επιτύχει αυτό και είναι ουσιαστικά απαραίτητη η απάντηση στην δεύτερη ερώτηση, το κατά πόσο είναι απαραίτητη για πολλά κράτη-μέλη, η απάντηση είναι όχι, διότι δεν έχουν βιομηχανία ανοιχτή θαλάσση και δεν ενδιαφέρονται. Δεν έχουν καμία ανάγκη για κάτι τέτοιο για τι υπόλοιπε χώρε που θέλουν, που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξη, μπορώ να δω κάποια πλέον εκτήματα. Αλλά η απόλυτη ομοφωνία από τη βιομηχανία και τι ενώσει και από τη Σκοτία και υπάρχει ομοφωνία επίσης και στην Νορβηγία ότι αυτό θα αποτελούσε βήμα προς τα πίσω έτσι όπως έχει συνταχθεί τόσο στους τύπο όσο και επί της ουσίας. Από λοιπόν άποψη Ηνωμένου Βασιλείου, Σκοτία και Νορβηγία, αυτό αποτελεί οπισθοχώρηση. Αυτό δεν ισχύει για την υπόλοιπη Ευρώπη, ίσω, αλλά θα χρειαστεί να είμαστε πιο ευέλικτοι στην ερμηνεία αυτού, του πακέτου μέτρων. Έχουμε τεράστια εμπειρογνωμοσύνη και φιλο... κοινέ φιλοδοξίε για το πώ θέλουμε να προχωρήσουμε. Θα αφιερώσουμε στη διάθεσή σα όλου του πόρου που έχουμε στη διάθεσή μα. Αλλά πραγματικά πρέπει να καταλήξουμε σε σωστή νομοθεσία. Αλλά η νομοθεσία είναι ενδιαφέρουσα εφόσον βελτιώνει την ασφαλεία του περιβάλλοντος και των εργαζομένων. Ε, συνάδελφος Βίνταλ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν να αναδείξω την ουσία του θέματο. Είναι αυτό το οποίο είπαν οι συνάδελφοι για την έκθεση του κ. Μπέλτ. Εγώ νομίζω ότι ακόμα η έκθεση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει παρουσιαστεί. Οπότε, εντάξει. Ε, φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ ε, τρομερό, <laughs> τρομερή ψήφο εμπιστοσύνη ε, που, που του αποδίδουν, αλλά είναι άλλο, άλλο τον άλλο το άλλο. Τώρα, επί του θέματος, νομίζω ότι αυτό ο κανονισμό παρουσιάζει κάποια θετικά, το ότι θέλει αυτός ο συντονισμό των, ε, των, των, των αποκρίσεων όταν υπάρχει κάποιο είδου κατάσταση ανάγκης ε, διασυνοριακή ή πιν. επίση συνεργασία μεταξύ των, των, των φορέων, των εταιριών, Όμω, έχουμε εδώ πέρα και κάποιε επικρίσει. Αυτέ οι επικρίσει δεν θα πρέπει να τι ξεχνάμε. Και επίση θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι όταν έρθει η ώρα ο εισηγητή να μα παρουσιάσει την έκθεσή του, να τα λάβει και αυτό υπόψη. Διότι, κοιτάξτε, ένα κανονισμό δεν είναι οδηγία. Είπαμε, είναι, καλύτερο, είναι καλύτερος από οδηγία, το οποίο αυτό είναι συζητήσιμο, αλλά ας, ας θεωρήσουμε ότι έχει αυτή, αυτό το, το, της άμεσης ε, εφαρμογής, ας το δεχθούμε. Όμως ε, αυτό είναι μια πρώτη άποψη, μια, μια, μια παραδοχή και άπαξ και θεωρήσουμε ότι έχουμε κανονισμό τότε από την άλλη μεριά ε, να δούμε το ότι κάποια κρατημέλη είναι ήδη πολύ προχωρημένο στον αφορά τη ρυθμισή του στην εθνική και με τον κανονισμό αυτό αυτά τα κρατημέλη εξαναγκάζονται, εξαναγκάζονται να προβούν σε κάποιες, σε κάποιες, σε κάποιες αλλαγές που δεν θα χρειαζόντουσαν. Ε, Επομένω αυτή η έκθεση ε, η οποία μας οδηγεί σε, ένα, σε μια τελική ρύθμιση, ένα τελικό αποτέλεσμα όσον αφορά τις οδηγίες, ε, θα πρέπει να καλύψει το ότι χρειάζεται να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Δηλαδή, αυτό το οποίο εδώ δεν το βρίσκω είναι το ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι ορισμοί που παίρνουν νερό που δεν είναι σαφείς τέλος όπως το άρθρο 2 και να γίνει επίσης και η διαφοροποίηση μεταξύ Εξόριξη ε, υψηλού κινδύνου και άλλες που δεν είναι υψηλού κινδύνου. Να μην θεωρήσουμε ότι όλα, όλα, όλα, όλα θα μας οδηγήσουν σε μια τραγωδία σαν τον κόλπο του Μεξικού. Αυτό ε, θα ήταν παράλογο. Άρα θα πρέπει η ρύθμιση να διακρίνεται από αναλογικότητα, δηλαδή εξασφάλιση, ε, προφύλαξη σε σχέση με τον κίνδυνο. Αυτό επίση και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αυτές τι προθεσμίε. Αν βάζουμε πάρα πολύ σύντομε προθεσμίε, τότε η προσαρμογή στου νέου κανόνε θα είναι τόσο, τόσο, τόσο επιβαρυντική για τις εταιρείε που θα έχουμε αντιπαραγωγικά αποτελέσματα όλα αυτά να τα έχουμε υπόψη. Και επομένω, πέραν όλων αυτών και εγώ ψηφίζω Μπέλετ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Χιζνάλφος Δεκαστήγιο. Όπως ε, είπατε και εσείς πρόεδρε, θα το ξανασυζητήσουμε. Θα υπάρξει χρόνος. Άρα σήμερα να μην συζητήσουμε ε, επί της ουσίας. Τα είπε και ο Πίτερ Σκίνερ ε, και έχουμε όλου αυτού του Άγγλου που ασχολούνται. Όμως ο εισηγητή δεν είναι Βρετανός, δεν είναι Βρετανός. Δεν έχουμε εδώ Βρετανού στην, στην ομάδα μας. Αμάν λέει, λέει. Αμάν, αλίμονο. Οπότε, να, τελικά ακούστηκε και η φωνή της, της Βρετανίας, γιατί δυστυχώς έλειπε τώρα. Θα πρέπει η συζήτηση για το αν θέλουμε διεκονίσμο να γίνει στο τέλος, στο τέλος. Και τώρα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ή στο περιεχόμενο. Συνέχεια τώρα να συζητούμε το αν θέλουμε το ένα ή το άλλο Φυσικά και τα επιχειρήματα που αναφέρονται είναι βάσιμα, όμως δεν ωφελεί τώρα αυτή η συζήτηση. Ας επικεντρώσουμε την προσοχή μα ή στο περιεχόμενο και η νομική φύση της ρύθμιση, αυτό είναι κανένα ας τα πούμε στο τέλος. Έτσι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Έτσι τώρα θα πάμε καλύτερα. Τώρα δεν μας βοηθάει καθόλου. Δεν προσθέτει τίποτα η συζήτηση για το νομοθετικό μέσο. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο βεβαίως τελικά να τοποθετηθεί. Θέλει το Κοινοβούλιο οδηγία ή κανονισμό. Ε, τότε θα ρίξουμε όλους μας το βάρος. Ευχαριστούμε Πιλάρ. Το λόγο έχει ο Ζαμπανέκ. Ζαμπανέκ. Παρακαλώ να μην μιλήσετε για πάνω από δύο λεπτά ώστε να δώσουμε ξανά το λόγο στην εισηγητή για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και όσους μίλησαν. Αφού έχω περιορισμένο χρόνο, δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε ο εισηγητής, πιστεύω ήταν καλά. Κάποια πράγματα υπάρχουν στην νομοθετική πρόταση από τη συζήτηση και τις ομιλίες των λοιπόν μελών καταλαβαίνω ότι έχουμε τον ίδιο σκοπό μας ε, απασχολεί το υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην Ευρώπη δεν θέλουμε να πάψουν να λειτουργούν αυτά που ήδη λειτουργούν σωστά σας διαβεβαιώ ότι εδώ έχουμε ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις απόψεις και τις ανησυχίες σας η πρόταση όπως ε, συντάχθηκε συντάχθηκε με μεγάλη προσοχή ώστε να μην δημιουργήσει προβλήματα. Επιλέξαμε κανονισμό για τους λόγους που αναφέρονται σε πάντοση τους έγγραφα. Θα το συζητήσουμε και περαιτέρω. Αντιλαμβάνομαι ωστόσο ότι ορισμένοι ενδιαφερόμενοι αντιτίθενται σε αυτό και ισχυρίζονται ότι ο κανονισμός θα είναι πολύ πιο δύσκολος ε, στην υλοποίηση. Εμείς παραμένουμε σε επαφή με ορισμένες από τις εθνικές αρχές που προωθούν αυτή την άποψη. Ακόμη δεν έχουμε ένα επιχείρημα το οποίο θα μπορέσει να στηρίξει αυτή την, ε, αυτόν τον ισχυρισμό. Έχουμε ακούσει διάφορες δηλώσεις όπως ακούσαμε σήμερα, αλλά όταν παίρνουμε σε λεπτομέρειες και ζητάμε μεγαλύτερη διαφάνεια, δεν τη βλέπουμε. Για παράδειγμα, δεν φαίνεται απαραίτητο για μας ε, όλες οι υποθέσεις ασφαλείας ε, να καταργηθούν, μπορούν απλά να τροποποιηθούν. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κανονισμός από αυτή την άποψη ε, αξίζει να θεωρηθεί ε, ε, ε, ικανός. Όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου έγιναν επικρίσεις, όσον αφορά τις μεθοδολογίες που εφαρμόζει η Κομισιόν, αλλά όταν συναντιόμαστε για να το συζητήσουμε με τους επικριτές των ενδιαφερομένων, έχουμε ήδη αξιολογήσει ομοτήμων, δεν ακούσαμε συγκεκριμένα λεπτομερή αντεπιχειρήματα που καθιστούν άκυρα τα στοιχεία της Κομισιόν. Έχουμε δει αξιόπιστα δεδομένα, αλλά τίποτα δεν ε, καθιστά αναξιά. Ε, μη ικανή τη δική μας ε, έκθεση. Το κατά πόσο τώρα ρέουν ή όχι από μόνα τους τα υγειοτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα. Έχουμε εξετάσει ολόκληρη την πετρελαϊκή βιομηχανία, όχι μόνο τη Βόρεια Θάλασσα. Δεν πρέπει να περιοριστούμε εκεί. Η εμπειρία λοιπόν Άλγεν είναι πολύ σημαντική. Σύμφωνο με όσου λένε ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα καθεστώτο που λειτουργεί και καλή απόκριση. Πήγε καλά, δεν χάθηκε καμία ζωή, δεν τραυματίστηκε κανεί και η περιβαλλοντική ζημιά ήταν πολύ περιορισμένη. Ωστόσο, θα θυμάστε όλοι ότι μετά από την εκένωση της εξέδρας για κάποιες ημέρες όλοι παρουσίαζαν διάφορες υποθέσεις γιατί άναψε και τι συνέβαινε και αν υπήρχε διαρροή και κανείς δεν είχε συγκεκριμένε απαντήσει για αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να προσέχουμε όταν ε, αξιολογούμε τις παρελθούσε εμπειρίες θέλουμε ακριβώ να αποφύγουμε καταστάσεις όπως αυτή που συνέβη πρόσφατα όπου φτάσαμε σε ένα σημείο που είδαμε ότι η νομοθεσία δεν είχε προβλέψει κάτι. Θέλουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη νομοθεσία η οποία θα μεριμνά για όλους τους κινδύνους και όχι μόνο για την υγεία και την ασφάλεια και για το περιβάλλον. Γενικά ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και ανυπομονώ να, εργαστούμε στενά γιατί να συνεργαστούμε στενά για τη βελτίωση της πρότασης. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι απαραίτητα και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ικανοποιητική νομοθεσία τελικά. Ωραία λοιπόν. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τους διερμηνείς για τα λίγα παραπάνω λεπτά που θα ε, διαρκεί η συνεδρίαση. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπελέτ λέγοντας το εξή Η παρουσίασή σας θα γίνει 11 Ιουλίου όπως συμφωνήθηκε όσον αφορά την ψηφοφορία για την εντολή διαπραγμάτευσης 9 Οκτωβρίου όπως είπατε εσείς ή μια ημερομηνία στην επόμενη συνεδρίαση 5 Νοεμβρίου αν δεν γίνει αυτή η συμφωνία με την ΕΜΒΗ. Ας αφήσουμε προς το παρόν το ημερολόγιο για αυτό το τελευταίο βήμα ε, σε εκκρεμότητα θα εξαρτηθεί από τις εργασίες των άλλων επιτροπών. Σας παρακαλώ να είστε σύντομος, θα μας κάνετε μια ολοκληρωμένη και ε, εξαιρετικά εξέπαινη παρουσίαση. Θα είμαι πολύ σύντομο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης εισηγητές και τους συναδέρφους για τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους ε, σχετικά. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, κυρία Πρόεδρε, θα θέλαμε να ε, μείνουμε στον Οκτώβριο, αλλά θα δούμε τελικά που θα καταλήξουμε. Θα έλεγα... Άκουσα όχι συνένεση, αλλά άκουσα παρόμοιες ε, παρατηρήσεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, την αρχή ο Ριπένων πληρώνει και τα υψηλά πρότυπα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τα πρότυπα που υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο ξέρουμε ότι υπάρχουν πολύ υψηλά πρότυπα. Το γνωρίζουμε αυτό λοιπόν. Χρειαζόμαστε επαρκή ευελιξία στο πλαίσιο των προτύπων αυτών όσον αφορά την νομοθεσία. Ε, ε, όσον αφορά το αν θα πρέπει να είναι οδηγία ή κανονισμός, Αναφερθήκατε στην ήδη προχωρημένη συζήτηση εντό του Συμβουλίου. Ίσως μπορέσουμε να βρούμε ένα δημιουργικό τρόπο να το λύσουμε αυτό. Αλλά συμφωνούμε με την Πιλάρο ότι δεν θα πρέπει να ε, παραλύσουμε λόγω της συζήτησης αυτής. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ουσία των πραγμάτων και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση που να παρέχει επαρκή ευελιξία. Άλλο σημείο που ήθελα να αναφέρω έχει να κάνει με το ρόλο της ΕΜΣΑ. Είναι σημαντικός ο ρόλος της ΕΜΣΑ. Θέλουμε να διευρύνουμε τον ρόλο της. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις, κυρία Ριβάζη, αναφερθήκατε στα, ε, στη χρήση των εσόδων των ε, επιχειρήσεων πετρελαίου και αερίου ε, για, για έρευνα και ανάπτυξη. Άλλο τρόπο θα ήταν ε, η ΕΜΣΑ να έχει περισσότερη ισχύ. Δεν ξέρω τι ε, γνώμη έχει η Επιτροπή. Είναι λεπτό το θέμα, αλλά πάση υπάρχει επιτάπητο τώρα η πρόταση αυτή. Επιτρέψτε μου κυρία Πρόεδρε να περιοριστώ σε αυτές τις παρατηρήσεις. Ε, Προσβλέπω στην επόμενη ε, ανταλλαγή απόψεων στις 11 Ιουλίου. Θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε την έκθεσή μας και θα έχουμε τότε τις πρώτες προτάσεις τροπολογιών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας για την εξαιρετική συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ τους διερμηνείς και θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 3 η ώρα. Ευχαριστώ.